Caras e caros colegas, eu devo eh, informar antes de mais eh, que estou, eh, presidir. συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι θα προεδρεύω εγώ εδώ, διότι δεν είναι εδώ ούτε ο πρόεδρος ούτε η Αντιπρόεδρε. Θα προσπαθήσω λοιπόν να κάνω ό,τι μπορώ προκειμένου οι εργασίες της Επιτροπής μας να μπορέσουν να διεξαχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όπως ε, γνωρίζετε, Η σημερινή συνεδρίαση θα διαρκέσει από τις 3 μέχρι τις 5 και μισή και αύριο το πρωί θα ξανασυνεχίσουμε στις 9 μέχρι και πάλι τις 5 και μισή το απόγευμα. Αύριο το πρωί θα έχουμε ψηφοφορίες. στις 9 και 4. Η συνεδρίαση ξεκινά στις 9, αλλά οι ψηφοφορίες ξεκινούν στις 9 και 4. Για να μην ε, χρονοτριβούμε άλλο όμως, να περάσουμε τώρα στην ημερήσια διάταξη. Σας έχει διανεμηθεί, νομίζω ότι μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη, δεν υπάρχουν παρατηρήσεις. Ωραία. Εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη και για σήμερα και για αύριο και περνάμε στο δεύτερο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Την έκθεση του συναδέλφου του κυρίου Λουίς Δεγκράντες Πασκουάλ ως προς τη ρήπανση από τα πλοία και θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις. Θα ήθελα λοιπόν να δώσουμε απευθείας το λόγο στον εισηγητή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως θα θυμάστε κυρίες και κύριοι, θα αναλύσουμε τις τροπολογίες που κατατέθησαν ε, στην ε, πρόταση τροποποίησης οδηγίας ε, για την ρήπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις Πρόκειται για την οδηγία 2005-667 ε, και είμαι εισηγητή αυτή τη έκθεση, όπω γνωρίζετε. Θα είμαι σύντομο, δεν θα σταθώ μόνο στι τροπολογίε, θα ήθελα να κάνω και μία αξιολόγηση για τα όσα παρουσίασαν οι συνάδελφοι και του ευχαριστώ ιδιαίτερα για το ενδιαφέρον του. Και θα εξάγω και κάποια συμπεράσματα, προσωπικά συμπεράσματα, ως προς τη βιωσιμότητα αυτής της πρότασης. Ε, πιστεύω ότι αν ενδιαφερθούμε όλοι, τόσο εμείς όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, θα μπορούσαμε να εκπληρώσουμε το όνειρό μα και να καταλήξουμε σε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Εμείς ως Επιτροπή Μεταφορών αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας λοιπόν και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα πάει η ψηφοφορία βάσει και αυτού του διαλόγου. Τώρα, για την πρόταση η πρόταση αυτή θέλει να πληρώσει το νομικό κενό που δημιουργήθηκε ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την απόφαση ε, πλαίσιο 2005-667 ΔΕΗ που ε, ολοκλήρωνε μια οδηγία άλλη και είχε σκοπό να πληρώσει ένα κενό που υπήρχε. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε ότι ο Ευρωπαίος νομοθέτης μπορεί να ε, αποφασίσει ως προς ποινικές κυρώσεις ε, σε θέματα πρώτου πυλώνα. Καταρχήν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι το μέτρο αυτό είναι απαραίτητο για να καταπολεμήσουμε τη ρήπανση από σκάφη και επίσης να πούμε ότι η λύση που εκφράζει, ε, που παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τα ελάχιστα όρια για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά κάτι πολύ συγκεκριμένο. Κατά την περίπτωσή μας τη ρήπανση που προέρχεται από σκάφη στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους πάντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να νομοθετεί, αλλά θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της πάντα και την ε, αρχή της επικουρικότητας. Θα πρέπει δηλαδή ε, τα κράτη-μέλη βάσει της αρχής της επικουρικότητας να αποφασίσουν ποια θα είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που θα ληφθούν. Εγώ εξ αρχής ε, έχω μια ανοιχτή θέση και δέχομαι τις προτάσεις των διαφορών πολιτικών ομάδων. Πρόθεσή μου εξ αρχής ήταν να έχουμε έναν ειλικρινή διάλογο με όλους όσους ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό. Ήθελα επίσης να δω και τι θα γίνει με τη γνωμοδότηση που ετοίμασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για το θέμα αυτό για να μπορέσουμε να έχουμε τις βασικές συνενέσεις που θα μας επιτρέψουν να έχουμε μια ποιοτική έκθεση. Αυτό και έκανα και ευχαριστώ και τα μέλη των ε, αρμοδίων επιτροπών ε, για τις ε, συνεισφορές τους και για τον ειλικρινή διάλογο ο οποίος ήταν καθόλου αφετικός για να μπορέσουμε να έχουμε συνένεση ως προς το θέμα αυτό. Επίσης μου φάνηκε ότι ήταν λογικό να μιλήσω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να έχουμε και κάποιες πρώτες εντυπώσεις από το Συμβούλιο. Λέω πρώτες εντυπώσεις διότι η νέα Προεδρία ε, πρέπει να καταλήξει και αυτή σε μία απόφαση και όπως μας είπε εδώ ο Υπουργός Μεταφορών τα θέματα των θαλάσσιων μεταφορών δεν είναι της ε, πείρας τους διότι η Τσεχία δεν έχει και τόσο πολύ θάλασσα. από αυτό το διάλογο και από τις εντυπώσεις που αποκόμισα από τους συναδέλφους είναι κάποιες τροπολογίες που παρουσιάστηκαν. Έχουμε 7 τροπολογίες που παρουσιάστηκαν από τους συναδέλφους Ρωτουέντο και Γεύνερ στην αρχική ε, έκθεση, μία τροπολογία που ενέκρινε η Επιτροπή Νομοθετικών Υποθέσεων, 7 ε, τροπολογίες που προκύπτουν από την γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και εγώ παρουσίασα δύο προφορικές τροπολογίες και αν δεν έχετε αντίρρηση ε, θεωρώ ότι είναι θετικές για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε τα όσα παρουσιάστηκαν στην έκθεση. Η μία είναι απλά μία βελτίωση στη διατύπωση, δεν έχει και μεγάλη σημασία. Και επίσης ε, έχω και ένα νέο εκτιμώντας το οποίο ε, δείχνει πόση σημασία δίνει ο εισηγητής ε, στα όσα κάνει ο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το τι γίνεται με την επανάληψη μικροαδικημάτων όταν φτάνουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ε, ναι μεν είμαστε θετικά διακείμενοι, αλλά υπάρχει και το εκτιμώντας το οποίο ε, εισαγάγει λίγο την αιτιολόγηση για το θέμα αυτό. Ως προς τις τροπολογίες που παρουσίασε ο κύριος Ορτουόντο, τον οποίο ευχαριστώ για τη βοήθειά του και για το διάλογο που είχαμε, παρουσίασε τέσσερις τροπολογίες βάσει και των παρατηρήσεων που έκανε και εδώ στην Επιτροπή όταν παρουσιάστηκε η εισήγηση την πρώτη φορά. Εγώ τις έλαβα υπόψη και θεωρώ ότι είναι θετικές διότι βελτιώνουν το κείμενο. Ο κύριος Ρωτουέντο δεν αλλάζει το κείμενο, ε, και θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι καλό. Και υπάρχει και μια συμβιβαστική τροπολογία με τον κύριο Ορτουόντορ για το σημείο 1α στο άρθρο 4, το οποίο καθορίζει ε, τις μικρές απορρίψεις, τα μικρά απόβλητα, τα οποία βελτιώνουν καλύτερα, ε, βελτιώνουν το κείμενο του εισηγητή. Σας το λέω με κάθε ειλικρίνη αυτό και επίσης είναι πάρα πολύ θετική η συνεισφορά του κύριου Ορτουόντου και λέει ότι αυτές ε, οι μικροαπορρίψεις είναι παράνομες. Αυτό στην έκθεσή μου δεν φαινόταν. Είναι αδικαιολόγητο να γίνεται κάτι τέτοιο γιατί κάνουμε διάκριση από τα, με βάση τα όσα έχουμε στη Σύμβαση Μαρπόλ. Επίσης αναφέρεται συγκεκριμένα το άρθρο 3 σημείο 1 για να καθορίσουμε το πεδίο εφαρμογής για, αυτές τις, ε, για αυτά τα απόβλητα, τα οποία είναι τελείως διαφορετικά από τα ε, μεγαλύτερες μορφές απόβλητα. Δεν μπορούμε δηλαδή να τα αποκλείσουμε από τη στενή έννοια της ε, απόφασης του δικαστηρίου. Υπάρχουν και κάποιες τροπολογίες οι οποίες είναι παρόμοιες με τις δικές μου, αλλά νομίζω ότι η διατύπωσή του είναι λίγο καλύτερη και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα μπορούσα να τις δεκτώ. Είναι οι 14 και οι 16, οι οποίες πληρούν τους στόχους του εισηγητή, αλλά παρουσιάζονται με καλύτερη διατύπωση. Και ο συνάδελφος Ορτουάντο απέσυρε την τροπολογία 15 γιατί θεωρεί ότι αυτό καλύπτεται από την τροπολογία 8 ε, του υποφαινόμενου. Τώρα, για τις τρεις ε, τροπολογίες του κυρίου Χούγνερ, ε, παρά το γεγονός ότι συμμερίζομαι τις ανησυχίες του, πιστεύω σοβαρά ότι για να συνεισφέρει θετικά αυτή τη στιγμή ε, θα είναι δύσκολο γιατί θα μπορούσαν να διακυβεύσουν ε, τα όσα έχουμε εμείς εδώ στην πρόταση. Φαίνεται ότι τα κράτη-μέλη μπόρεσαν να έχουν μια συνένεση ω προς τις βασικέ έννοιε και αν κάνουμε εμεί αλλαγέ τώρα μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Το δέχεται και ο συνάδελφο Χέμπνερ αυτό στη διμερή συνάντηση που κάναμε αυτό, γι' αυτό και ακριβώ δέχτηκε να αποσύρει δύο από τι τροπολογίε πιο συγκεκριμένα τι τροπολογίε 17 και 18. Ε, θεωρώ ότι είναι θετική όμως η τροπολογία, συγγνώμη, αποσύρει τις τροπολογίες 17 και 19, θεωρώ ότι είναι θετική η τροπολογία 18 του κυρίου Έμπνερ και θεωρώ ότι είναι θετικά τα στοιχεία διότι έχουν ένα επιπρόσθετο έφυλ, όφελος τα όσα προτείνουμε διότι απαντά στα ερωτήματα που θέτουμε εμείς ε, συνεχώς. Ποιο αξιολογεί τι συνέπειε τη ρήπανση που προκύπτει. Και επίση θα ήθελα να σα υποθυμίσω και τον κανονισμό που εγκρίναμε πριν από δύο χρόνια, στα οποία ήμουν και πάλι συγητή και ζητούσαμε από την ΕΜΣΑ, στην Υπηρεσία για την Ναυτιλιακή Ασφάλεια, ασφάλεια να λάβει υπόψη ε, το θέμα της ρήπανσης από σκάφη στα ευρωπαϊκά ύδατα και δεσμευόντουσαν να έχουν μία υπηρεσία εικόνων δορυφορικών για να μπορέσουμε να έχουμε στοιχεία για τη ρήπανση και να μπορούμε να εντοπίσουμε και ποια είναι τα υπεύθυνα σκάφη. Με την πρόταση που γίνεται από το συνάδελφο Έμπνερ, το να έχουμε δηλαδή ένα μέσο το οποίο θα αναλύει τα στοιχεία και θα δίνει τα δεδομένα σε βιολογικό, χημικό και φυσικό επίπεδο, πιστεύω ότι καλύπτεται αυτό ο στόχο, ο οποίο προέκυψε από την έκθεση του 2007. Δεν πρόκειται για κάτι λοιπόν ε, καινοφανέ είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως αποτελεί καθήκον της ΕΜΣΑΝ και το είχαμε ζητήσει στην ετήσια έκθεση για τη χρηματοδότησή του. Τώρα, για τις ε, τροπολογίες της Επιτροπής Νομικών ε, Υποθέσεων. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλές διότι διασφαλίζουν μεγαλύτερη συνοχή και νομική ασφάλεια και έχουν δύο νομοθετικές προτάσεις που έχουν δύο βασικά στοιχεία. Ε, τα ίδια είχαμε και στο πακέτο ΕΡΙΚΑ 3, το οποίο εκκρεμεί ω προ την έγκρισή του, όπω ξέρετε όλοι, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα βρίσκεται τον επόμενο μήνα στι προτάσει. Ε, Η τελευταία φράση του κειμένου, δηλαδή την εισαγωγή κοινικών πυρώσεων για οποιαδήποτε ε, παράνομη απόρριψη, νομίζω ότι δεν είναι αποδεκτή, διότι αναφέρεται αποκλειστικά σε όλες τις περιπτώσεις που πληρούν τις ε, προϋποθέσεις που ε, καλύπτει η απόφαση του δικαστηρίου. Οι επτά τροπολογίες που παρουσιάστηκαν βρίσκουν σύμφωνο τον εισηγητή σε πέντε τροπολογίες, τις 1, 2, 3, 4 και 5, οι οποίες συνεισφέρουν και βελτιώνουν τη διατύπωση του κειμένου και βοηθούν και την καλύτερη κατανόηση. Όμως ε, είμαι καθόλου αντίθετος και το λέω και στον ενδιαφερόμενο για την ε, τροπολογία 6 και ζητώ και πάλι την υποστήριξή σας. Ε, θα ήθελα να απορριφθεί αυτή η τροπολογία διότι καλύπτει, διαγράφει συγγνώμη το θέμα της σοβαρότητας και θεωρείται ως ποινικό οτιδήποτε προκύπτει από συγκεκριμένη ευθύνη παρά το γεγονός ότι δεν το επιτρέπει η απόφαση του δικαστηρίου. Υπάρχουν συγκεκριμένα όρια τα οποία καθορίζουν η απόφαση του δικαστηρίου, αλλά ο κανονισμός αναφέρεται και σε ποινικέ κυρώσει όταν πληρούνται συγκεκριμένε ε, προϋποθέσεις, όταν υπάρχει σοβαρή αμέλεια παραδείγματι. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα στοιχεία αυτά, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τα συζητάμε άλλο εδώ. Τώρα, για τι προφορικέ τροπολογίε του εισηγητή. Ζητώ και την κατανόησή σα ε, για το θέμα αυτό, γιατί θέλω να παρουσιάσω δύο τροποφορικέ τροπολογίε. Η πρώτη έχει ω στόχο να βελτιώσουμε τη διατύπωση της, ε, ε, του σημείου 4, του άρθρου 4. Είναι καθαρά θέμα διατύπωση και στυλ. Και η επόμενη, όπω σα εξήγησα, είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι έχουμε πλήρη. Ε, συνάφεια με τα όσα παρουσίασε ο εισηγητής. Έχουμε τις μικροπαραβάσεις ε, όταν πληρούνται ε, προϋποθέσεις αμέλειας ή δόλου. Αυτά λοιπόν ε, ως προς τις τροπολογίες, αυτή την έννοια έχει η εκθεσή μου και αυτή είναι η θέση που θα ήθελα να σας παρουσιάσω και θα ήθελα να σας ζητήσω κύριε Πρόεδρε την κατανόησή σας, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση τώρα και ζητώ συγγνώμη αν μακρηγόρησα. Ευχαριστώ πολύ. E σας ευχαριστώ κύριε Πασκάλ. Να δώσω το λόγο στην κυρία από Η κυρία Μιγγέλες Ράμος. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να παρέμβω για να πω ότι υποστηρίζω τις θέσεις ε, του εισηγητή, του κύριου Ντεγκράντες Πασκουάλ, διότι όπως ε, είπε και ο ίδιος, η έκθεση αυτή, την οποία συζητάμε σήμερα, πληρεί τις αρχές ε, των οποίων αποτέλεσε έμπευση. Καταρχήν υπάρχει μια ισορροπημένη ε, σύνθεση των δύο αποφάσεων που έχουμε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ταυτόχρονα υπάρχει και η ανάγκη να εναρμονιστεί και να ομογενοποιηθεί η Σύμβαση Μαρπόλ για όλα τα κράτη-μέλη ε, μετά από τα προβλήματα που προέκυψαν λόγω αυτής της κατάστασης και επίσης όπως το επεσήμανε και ο ίδιος ο εισηγητής και νομίζω ότι αυτό είναι αυτό το οποίο επέμενε περισσότερο και είναι και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η διάκριση μεταξύ διοικητικών κυρώσεων για να επιβάλλονται κυρώσεις σε μικροπαραβάσεις, σε μικροαπορρίψεις και σε μεγαλύτερες κυρώσεις για τις ε, περιπτώσεις τις οποίες ε, η ζημία που προκαλείται είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ αυτών των δύο συμπεριφορών, αυτών των δύο θεμάτων. Και γι' αυτό ακριβώς μου φαίνεται ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι σε αυτή την έκθεση, και νομίζω ότι το επέτυχε αυτό ο εισηγητής με την ε, διατύπωση που παρουσιάζει, ότι είναι σημαντική η ανάγκη να θεωρείται ποινικό αδίκημα το να έχουμε κατ' επανάληψη μικροπαραβάσεις. Διότι αν κάποιο συνεχώς επαναλαμβάνει αυτές τις μικροπαραβάσεις, ε, σημαίνει ότι θα έχουμε ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη ρήπανση. Και επίσης ε, διότι σε αυτές τις συμπεριφορές, ε, σε πολλές περιπτώσεις, και αυτό το παρατηρούμε άλλωστε και στην ζωή μας καθημερινά, υπάρχει πρόθεση ή υπάρχει και αμέλεια, σοβαρή αμέλεια. Και δικαίως λοιπόν αυτός ο κανόνας τον οποίο θέλουμε να εγκρίνουμε εδώ έχει αυτό το πλεονέκτημα. Δεν ε, κάνει διάκριση μεταξύ αυτών των δύο συμπεριφερών. Θα ήθελα να πω στον κύριο Ντεγκράντε ότι σε γενικέ γραμμέ η πολιτική μου ομάδα συμφωνεί με τι ε, θέσει σα και συμφωνεί επίση και με τον κατάλογο των ψηφοφοριών. Θα ήθελα μόνο να μου κάνει ένα σχόλιο για μία από τις δικές του τροπολογίες. Η τροπολογία που αλλάζει την ε, περίοδο μεταφοράς αυτής της ε, πρότασης οδηγίας, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ε, ένα διάστημα 6 μηνών και ο εισηγητής προτείνει 12 μήνες. Επειδή σε γενικές γραμμές τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι προετοιμασμένα για να εφαρμόσουν αυτή την οδηγία το συντομότερο δυνατόν ε, αυτή τη στιγμή εγκριθεί. Θα ήθελα να ξέρω με ποιο τρόπο δικαιολογεί ο κ. Δεγκράντες Πασκουάλ το γεγονός ότι σε αυτή την τροπολογία ε, φαίνεται να αλλάζει την προθεσμία. Ποια γραμμή θα ακολουθήσουμε εμείς, τους 6 μήνες που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τους 12 μήνες που προτείνετε εσείς στην τροπολογία σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Λίστεμπεργκ έχει το λόγο. Κυρία Λίστεμπεργκ, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή. Είναι πολύ σύμφωτο το θέμα αυτό. Για ένα λόγο. Γιατί στον τομέα αυτόν βρισκόμαστε στα πρώιμα στάδια, αν θέλετε, οπότε δεν μπορούμε συστηματικά και αποτελεσματικά να αναπτύξουμε αξιόπιστα συστήματα σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό. Και δυστυχώς η απόφαση του δικαστηρίου δεν μας δίνει την απαραίτητη ευελιξία για να μπορέσουμε να εισάγουμε αποτελεσματικά μέτρα. Είμαι θετική σε ό,τι αφορά την προσέγγιση αναφορικά με τις επαναλαμβανόμενες απορρίψεις και, μικρής, και μικρών ποσοτήτων ότι θα πρέπει αυτό να οδηγεί σε ποινές γιατί μιλάμε για μεγάλες ζημιές, προκαλούνται μεγάλες ζημιές. Αυτό πολύ απλά θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το εξή ότι η δίωξη των αξιόπινων αυτών πράξεων είναι κάτι το πολυσύνθετο. Και να διαπιστώσουμε ποιος είναι ο υπεύθυνο να αποδώσουμε την ευθύνη στη συνέχεια. Αυτό απαιτεί όχι μόνο χημικές αναλύσεις, αλλά και πολυσύνθετες νομικές διαδικασίες στον τομέα αυτό. Ακριβώς λοιπόν επειδή είναι τόσο σημαντικές οι ζημιές που προκύπτουν, εγώ θα πίστευα και θα ήθελα να παρακαλέσω τον εισηγητή να το βάλει αυτό σε ένα εκτιμώντας, να το κοιτάξει μάλλον αυτό σε ό,τι αφορά την τελευταία πρόταση ενός εκτιμώντας, γιατί λέει ότι δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει ενδεχόμενες ποινικέ κυρώσεις, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το εξή. Ξέρω ότι τα κράτη-μέλη παλεύουν και αγωνίζονται κατά την εισαγωγή ποινικών κυρώσεων από ευρωπαϊκής πλευράς. Γνωρίζω πώς έχει η συζήτηση και τι συζητιέται και στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων κυρίως και με τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Να πω όμως το εξή ότι σε κάποιους τομείς, χωρίς τον μηχανισμό αυτών των μηνικών κυρώσεων, δεν πρόκειται να τα βγάλουμε πέρα. Σας το λέω ξεκάθαρα. Δεν θα μπορέσουμε να εισάγουμε αποτελεσματικά μέτρα κατά επανειλημμένων τέτοιων απορρίψεων κατά συρροή, δεν θα μπορέσουμε να εισάγουμε αποτελεσματικά μέτρα χωρίς αυτή την πτυχή. Γιατί πολύ απλά θα συνεχιστεί η ήδη φυστάμενη πρακτική. Γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχουν σημαντικές συνέπειες σήμερα. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε και αυτό να μπει σε ένα εκτιμόντο, σε μια τελογική σκέψη, να μην έχει άμεση εφαρμογή δηλαδή. γιατί νομίζω ότι στο θέμα αυτό θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αντιμετωπίζουμε συστηματικά περιβαλλοντικά εγκλήματα. Και είναι νομίζω καταφανή τα παραδείγματα. Και είναι δύσκολο να επανορθωθούν οι ζημιές αυτές. Η ζημιά για τον τουρισμό, η ζημιά για την αλληλεία και για πολλούς άλλους κλάδους. Νομίζω λοιπόν ότι το θέμα αυτό θα μας απασχολήσει πολύ στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν και καλό τον εισηγητή να το σκεφτεί το θέμα αυτό, γιατί δεν πρόκειται και για κάτι που είναι άμεσα εφαρμόσιμο, θέτει απλά μία μελλοντική προοπτική. Να το σκεφτεί. Να σκεφτεί μήπως θα έπρεπε να συμπεριληφθεί και αυτή η προσέγγιση. Γιατί πρόκειται για μόνιμες ε, ζημιές στο περιβάλλον βλάβες, οι οποίες δεν μπορούν να επανορθούν. Και ουσιαστικά με τις διοικητικές ε, ποινές που επιβάλλονται σήμερα δεν πετυχαίνουμε σπουδαία πράγματα, γιατί δεν τις παίρνουν στο σοβαρά όσοι κάνουν τα εγκλήματα αυτά. Και φυσικά τίθεται και θέμα διαφορετικών συστημάτων στα κράτη-μέλη και διαφορετικών πραγματικότητων. Αν μας δυσκολεύουν λοιπόν τόσο πολύ οι ποινές και το θέμα των ποινών, θα πρέπει να φροντίσουμε τουλάχιστον όταν βρίσκουμε τον υπεύθυνο, όταν βρίσκουμε τον υπέτειο, να έχουμε στη διάθεσή μας επαρκή μέσα, επαρκή κυρώσεις, γιατί μετωπίζουμε τεράστια προβλήματα. Δεν πρέπει να τα υποτιμούμε τα προβλήματα αυτά και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι θέμα μόνο που αφορά την ε, ναυτιλία, αλλά Πρόκειται για κάτι που το οποίο θα επηρεάσει στο μέλλον όλο και πιο πολύ τους εσωτερικούς πλατούς διαδρόμους. Γενικώ πώς? Δυστυχώς δεν μπορούμε να εργαστούμε πραγματικά αποτελεσματικά λόγω της ε, δικαστικής απόφασης, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να εξαντλήσουμε ό,τι μέσα έχουμε στη διάθεσή μας για να αποστείλουμε και ένα μήνυμα προς το Συμβούλιο. για τα συστηματικά αυτά ε, επιχειρήματα που έχουμε και για το ότι θα ανεχτούμε τέτοιες πράξεις. Ευχαριστούμε πολύ. Συμφωνώ με την προηγούμενη ομιλήτρια και εμεί θα θέλαμε να είχαμε στα μέσα, στην διάθεσή μας ε, ποινικά μέσα, αλλά συμφωνώ με τον εισηγητή μας. Δεν έχει οποιοδήποτε λόγο να υπάρχει μια τέτοια έκκληση σε μια αιτιολογική σκέψη. Πρόκειται για μια συζήτηση επί της αρχής που θα πρέπει να γίνει με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Να το δούμε και πέρα από τις συνθήκες Λισαβόνας. Πρόκειται για ένα θέμα επί της αρχής λοιπόν, βλέποντας ότι τα εθνικά κράτη δεν δημιουργούν το απαραίτητο ποινικό δίκαιο, όταν δεν υπάρχει λοιπόν αυτό το απαραίτητο ποινικό δίκαιο σε επίπεδο εθνικού κράτου μέλου, θα πρέπει να υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν υπάρχει όμω σήμερα αυτή η αρμοδιότητα, αυτό το βλέπουμε. Και έτσι όπως έχει σήμερα η έκθεση, τι λέμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε διοικητικό επίπεδο είναι πραγματικά κάτι σημαντικό, είναι σημαντικό όπλο στα χέρια μας. Θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε στο έπακρον και με πείθουν όλες ε, οι τροπολογίες που έχουν υποβληθεί από τις διάφορες επιτροπές. Θα πρέπει τουλάχιστον να ψηφίσουμε αυτό το μέσο προκειμένου τουλάχιστον τα μέσα που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας να τα χρησιμοποιήσουμε. Και κατά τη συζήτηση για την έκθεση, φυσικά και θα πρέπει να θίξουμε το θέμα αυτό. Μήπω εξ δηλαδή θα πρέπει να αλλάξουμε την προσέγγιση μα. Όντω δηλαδή, όπου υπάρχει πρόβλημα όχι μόνο σε ό,τι αφορά το περιβάλλον αλλά και σε άλλους τομέες όπου τα κράτη-μέλη δεν ανταποκρίνονται επαρκώς θα πρέπει ίσως σε ποινικό επίπεδο να εισαχθούν ευρωπαϊκά μέτρα. Χαίρομαι που συμφωνούν όλες οι ομάδες και νομίζω ότι θα πρέπει αύριο να υπερψηφίσουμε όλη την έκθεση του συναδέλφου για να πούμε, να δώσουμε ένα ε, μήνυμα προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι θέλουμε να υπάρξει κάποια ανταπόκριση. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τι είχαν να πούνε οι συνάδελφοι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο και στη συνέχεια μπορεί να καταλήξει συμπεράσματα ο Παρακαλώ. Euh, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Δεν θα ήθελα καταρχάς να επαναλάβω τα όσα ήδη σας είπα στην προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής σας, όταν πρωτοπήρα το λόγο για να αντιδράσω στην έκθεση και στις τροπολογίες του κυρίου Ντεγκράντες Πασκουάλ, να κάνω απλώ δύο παρατηρήσεις. Να σε επενθυμίσω πρώτον ότι προσπαθούμε εδώ πέρα να εργαστούμε βάσει του υφιστάμενου δικαίου και προσπαθούμε να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες που μας δίνονται για την τροποποίηση της υφιστάμενης οδηγίας, προκειμένου να καταφέρουμε δηλαδή να συμμορφωθούμε με τις αποφάσεις του 10, κρατώντας όμως αν θέλετε, το εφιστάμενο σύστημα το οποίο είχε προτείνει το Συμβούλιο, δηλαδή να έχουμε μία οδηγία και μία απόφαση πλαίσιο η οποία έχει να κάνει με τις ποινικέ κυρώσεις. Θα θυμάστε το δικαστήριο είπε ότι αν ο νομοθέτης κρίνει αναγκαίο να κάνει μια τροποποίηση, τότε στα πλαίσια του πρώτου πυλώνα μπορούμε να έχουμε ποινικέ κυρώσεις έτσι ώστε να πετύχουμε τους στόχους του κοινοτικού δικαίου. Σε αυτό προσβλέπουμε, στο εγχείρημα αυτό, χωρίς όμως να έχουμε την πρόθεση να τροποποιήσουμε την ουσία των κοινοτικών διατάξεων. Πρώτον αυτών. Δεύτερον, το επενθύμησε αυτό και στην προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής σας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα ήταν αρκετά συντηρητική, συγκρατημένη όσον αφορά τις λεγόμενες ελάσσονες απορρίψεις. Πώς μπορούμε να μιλάμε για ρήπανση η οποία ουσιαστικά δεν επηρεάζει την ποιότητα των υδάτων καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να κάνουμε μια τέτοια εκτίμηση και αξιολόγηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, βλέπουμε ότι μέσω τροπολογιών έχουμε το νέο αυτό στοιχείο, μιλάμε για ελάσσονες απορρίψεις, καταλαβαίνω ότι απορρέει η έννοια αυτή από την απόφαση πλαίσιο, θα πρέπει να καταλάβουμε όμως ότι η νέα αυτή συμπερίληψη έχει και κάποιες επιπτώσεις. Άκουσα τον εισηγητή, την κυρία Λιχτεμπέργκερ επίσης, καθώς επίσης και την κυρία Μιγγέλες Ράμος, οι επανειλημμένες ελάσσονες απορρίψεις προκαλούν ένα πρόβλημα, δημιουργούν κάποιες δυσκολίες. Ε, εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν και κάποιες ακόμα διαδικαστικές δυσκολίες. Πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε τον επαναληπτικό χαρακτήρα αυτών των απορρίψεων. Πότε ξεκινά ο επαναληπτικός χαρακτήρας. Μέχρι ποιο αριθμό μπορούμε να φτάσουμε. Σε ποιο βαθμό. Και αυτό πρέπει να το αξιολογήσουμε. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι ε, οι τροπολογίες του κυρίου Ορτουόντο είναι ουσιαστικά μία επαναδιατύπωση των όσων προτείνει ο κύριος Ντεγκράντες Πασκουάλη. Θα ήθελα λοιπόν να αφαιρθώ σε αυτές. Υπάρχει όμως μία τροπολογία η οποία μου δημιουργεί πρόβλημα, τροπολογία 18 συγκεκριμένα. Η τροπολογία αυτή ουσιαστικά που αναφέρεται στις τρεις προηγούμενες τροπολογίες του κυρίου Έμπνερ. Δεν θα ήθελα να αξιολογήσω την τροπολογία αυτή καθ' αυτή. Θα ήθελα απλώς να σας πω ότι αν διατηρήσουμε αυτή την τροπολογία, τότε καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου δεν θα καταφέρουμε να εφαρμόσουμε το υφιστάμενο δίκαιο και αυτό καταλαβαίνετε ότι προκαλεί μια δυσκολία. Τώρα, όσον αφορά τις τροπολογίες Επιτροπής Περιβάλλοντος, όπως το είπε και ο εισηγητής, έτσι και εγώ θα ήθελα να πω ότι ε, σημαντικό πρόβλημα προκαλεί κατά τη γνώμη μου η τροπολογία υπαριθμών 6 που έχει ως στόχο να τροποποιήσει με τρόπο ιδιαίτερα ισχυρό το ηθικό στοιχείο το οποίο βρίσκεται στη βάση της παράβασης. Πιστεύω εδώ πέρα ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί και πάλι το εφιστάμενο δίκαιο και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στην εφαρμογή των όσων λέει η τροπολογία αυτή. Αυτή είναι τουλάχιστον η άποψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος, να αναφερθώ στι τροπολογίε της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και συγκεκριμένα στο σημείο 3α του άρθρου 4 Πιστεύω ότι ε, μπορούμε να αποδεχτούμε εμεί εξ ονόμου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ε, προτινόμενη αυτή τροπολογία. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. ευχαριστώ. Να δώσω τον λόγο στον εισηγητή για να κλείσει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ε, συναδέλφους και συναδέλφους που παρενέβησαν για να εκφράσουν την άποψή τους. Να ξεκινήσω με την κυρία Μικέλες Ράμος, τη συμπατριωτήσά μου. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την θετική στάση που έχετε ως προς το σύνολο της, της έκθεσής μου. Νομίζω ότι το πνεύμα τη έκθεσή μου το έχουν κατανοήσει όλο, όλοι, παρά το γεγονό ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορέ στο ένα ή στο άλλο σημείο. Και φαίνεται την κυρία Μικέλε Ράμο να την ανησυχεί κάτι που εμένα μου φαίνεται όχι και τόσο σημαντικό. Να γίνω πιο σαφής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 6 μήνε εγώ 12. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αίσθηση από πλευρά του Συμβουλίου και από πλευρά κάποιων συναδέλφων που προτείνει να φτάσουμε μέχρι και τους 24 μήνες, ούτε καν 12, 24 και περισσότερους. Ε, γιατί υπάρχει μια αίσθηση ότι μπορούν να κυλήσουν λίγο περισσότερο τα πράγματα. Ε, αλλά εμείς κάνουμε μια πρόταση για να έχουμε μια κάποια ισορροπία. Και αυτή είναι η πρότασή μου. Και αν είναι αλήθεια το όσα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτό το θέμα ούτως ή άλλως ε, το έχουμε εξετάσει και ξέρουμε ότι μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα, τότε ε, θα μπορούσαμε να δεχτούμε και τη δική τους ε, πρόταση. Το, οι 12 μήνε δεν είναι μια προθεσμία που δίνει ένα, μια ιδέα ότι μπορεί να καθυστερήσουν και άλλα τα πράγματα και να παρακολύσουμε τις καταστάσει Οι άλλες ε, προτάσεις που είχαμε ε, νομίζω ότι οδηγούσαν σε καθυστερήσεις. Αυτό λοιπόν, σε καμία περίπτωση να ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο, νόμιζα ότι αυτή ήταν η συνένεση ανάλογα ανάμεσα στις προτάσεις που είχα. Ήθελα δηλαδή να συγκεράσω όλες τις απόψεις. Σας ευχαριστώ παρόλα αυτά κυρία Μιγγέλα Στράμος για τόσα κάνετε. Κυρία Λίχτεμπεργκερ, προσπάθησα να μιλήσω μαζί σας. Έχουμε συζητήσει διαμακρών για το θέμα αυτό. Είστε ένα αξιότιμο μέλος της ε, Επιτροπής μας, εγνωσμένου κύρους και άλλωστε είστε και η συντάκτρια της νομοδότησης της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Υπάρχει και μια σύγκρουση αρμοδιοτήτων και αποφασίστηκε από εκεί ότι θα λάβουμε εμείς το ε, θα αναλάβουμε εμείς το θέμα. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που ήσασταν τόσο δεκτικοί. Δεν θέλω να σας διασκεδάσω τις αμφιβολίες, διότι το θέμα αυτό έχει πάρα πολλές αμφιβολίες. Πώς μπορούμε να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ Ελλάσσων και μίζωνων θεμάτων δεν ξέρω. Η τροπολογία του κυρίου Έμπνερ. Αύριο εγώ θα μιλήσω με τον υπεύθυνο του ε, Οργανισμού για την Θαλάσσια Ασφάλεια και θα του τα θέσω αυτά τα θέματα. Διότι καλό θα ήταν να είναι και αποτελεσματικοί ως προς τα καθήκοντά του αυτή του οργανισμού, αλλά εγώ δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει τέτοια δυνατότητα με δραστικό τρόπο. Τώρα, υπάρχουν οι εξή ανησυχίε. Πρώτον, γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλησε ποτέ να κάνει διάκριση μεταξύ ελάσσονων θεαμάτων. Αλλά υπάρχει και το Συμβούλιο στη μέση και το Συμβούλιο θα πρέπει να εκφράσει την άποψή του και το Συμβούλιο ανησυχεί ότι ε, ε, αυτή η απόφαση από πλευράς νομολογίας και όχι μέσω αλλαγής της ε, συνθήκης ε, και το γεγονό ότι δίνονται δυνατότητες σε ποινικές κυρώσεις στον πρώτο πυλώνα άνοιγε πάρα πολύ τις δυνατότητες. Γι' αυτό ακριβώ και θέλησα να κάνω τη διάκριση μεταξύ των ελάχιστων θεμάτων και των θεμάτων ε, τα οποία θεωρούνται πιο σοβαρά. Και δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να ε, ε, μη λάβουμε υπόψη μας αυτό το θέμα, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με αποφάσεις στο δικαστήριο. Αυτό μου δείχνει και η πείρα μου ως νομικός. Και δεν πρέπει να εκμεταλλευτούμε την, την κατάσταση με αρνητικό τρόπο. Μπορούμε να φτάσουμε μέχρι ένα σημείο, αλλά όχι να το παρατραβήξουμε. Θα πρέπει να φτάσουμε μέχρι τις αρμοδιότητές μας και να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχει το θέμα της επικουρικότητας. Είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα ε, σοβαρό και μέχρι εκεί μπορούμε να φτάσουμε. Εγώ συμμερίζομαι λοιπόν τις ανησυχίες σας για αυτές τις δυσκολίες, αλλά δεν μπορούμε να υπερβούμε τα σκαμμένα. Επειδή κάνουμε διάκριση σε ελάσσον και πιο σοβαρές ε, απορρίψει, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και ένα θέμα το οποίο είναι γεγονό και είναι πολύ σημαντικό. Το γεγονό ότι οι τέτοιε συμπεριφορέ σε μικροαπορρίψει είναι ούτω ή άλλω ε, ε συμπεριφορέ που είναι πάρα πολύ σοβαρή αμέλεια και είναι επαναλαμβανόμενε και πολλέ φορέ οδηγούν σε σοβαρή ρήπανση. Πρόκειται λοιπόν δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα και δεν έχουν ε, παρά μόνο διοικητικέ κυρώσει, ουσιαστικά ε, απλά και μόνο θα πληρώνουν τα πρόστιμα. Εμεί θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη ρήπανση με δραστικό τρόπο και αυτή είναι η ίδια ανησυχία με αυτή που έχετε κι εσεί. Τελικά θα έχουμε αποτελέσματα με αυτόν τον κανόνα. Όχι, κατά πάσα πιθανότητα όχι. Αυτό που μα δίνει τη δυνατότητα όμω να κάνουμε είναι να τηρήσουμε τους στενούς όρους της απόφασης αλλά όχι να πάμε πολύ παραπέρα. Γι' αυτό λοιπόν σας ζητώ προσοχή και ε, πολύ υπομονή για να μπορέσουμε να καταλήξουμε εμείς σε συνένεση, να μιλήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να μιλήσουμε και το Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν Τσεχική Προεδρία λέει ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει θαλάσσια θέματα τόσο καλά. Ας εκμεταλλευτούμε τη δυνατότητα για να έχουμε και μια γενικευμένη συνένεση η Επιτροπή Μεταφορών αυτό πρέπει να κάνει, θα πρέπει να θέσει ένα όριο και από εκεί και πέρα ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ας περάσουμε τώρα στο τρίτο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Θα συζητήσουμε για τη δημιουργία του κοινού αεροπορικού χώρου με το Ισραήλ. Δίνω ευθύ αμέσω ε, το λόγο στον εισηγητή, Ρωμανιόλη. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Κύριοι συνάδελφοι, σε προηγούμενες συνεδρίες σας παρουσίασα την έκθεση και μιλάμε για μια έκθεση προοπτικών πολύ σημαντικών για τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η στρατηγική τους ανάπτυξη Μα βοηθά να διαπιστώσουμε ότι θα έχουμε πολλά ωφέλη και όχι μόνο οικονομικά για όλες τις πλευρές, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το Ισραήλ σίγουρα, αλλά ελπίζω και για την Παλαιστίνη. Στην ε, παράγραφο 1 προτάθηκαν κάποιε τροπολογίε από του αδέλφου τη ΓΚΟΕ. Αυτού δεν μπορώ να τι δεχτώ σε καμία περίπτωση, διότι αφενό ε, ε, παρακολύουμε την ανάπτυξη τη συνεργασία με όλη τη Μέση Ανατολή και με το Ισραήλ αλλά και με την Παλαιστίνη και ουσιαστικά κατά την άποψή μου εισάγεται και μία καθυστερημένη βεβιασμένη καθυστέρηση η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα βοηθήσει τη λύση της ε, αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο χωρών. Εγώ δεν θα ήθελα να δω ε, το θέμα της διατύπωσης που χρησιμοποιείται στο εκτιμώντας. Ε, θεωρώ ότι υπάρχει πολιτική δυνατότητα να εκφράσουμε κάτι τέτοιο, αλλά θα ήθελα να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι η ανταλλαγή εμπορευμάτων, ανθρώπων, ε, υπηρεσιών, οτιδήποτε άλλο, η ελευθερία δηλαδή, οτιδήποτε, οποιοδήποτε παράγοντα που επιτρέπει την ελεύθερη μετακίνηση, την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων, ήταν πάρα πολύ σημαντικές ε, και η παραβίασή τους ήταν αποτέλεσμα πολλών απολυταρχικών καθεστώτων. Για να μην ξεχνάμε και τα πρώην κομμουνιστικά κράτη της Σοβιετικής Ένωσης κλπ. Υπάρχει και μια Ιταλική παροιμία που λέει ορισμένες φορές κάνει μεγαλύτερη ζημιά το βαμβάκι παρά το σπαθί. καλύτερο θα ήταν να μην έχουμε ελεύθερη μετακίνηση παρά να έχουμε αυτή την βεβαιασμένη πάυση των εργασιών. Το να δίνουμε την έγκριση στο Ισραήλ για κάτι τέτοιο νομίζω επαναλαμβάνω ότι δίνει και στην Παλαιστίνη τη δυνατότητα για ανταλλαγέ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και με τις ε, υπόλοιπε χώρες του κόσμου. Αν θέλαμε για παράδειγμα να κατασκευάσουμε ένα αεροδρόμιο στη Γάζα και κλείναμε αυτό που θα είχαμε στο Ισραήλ τότε καταλαβαίνω ότι οποιαδήποτε παρατήρηση θα μπορούσε να έχει μια διαφορετικό νόημα και θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Επειδή όμω δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι δίνεται δυνατότητα να αναπτύξουμε άλλον ένα αέριο χώρο από αυτόν που προτείνεται και δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι το να διακοπούν οι διαπραγματεύσει με το Ισραήλ δεν θα βοηθήσει κανένα από τα συμβαλόμενα μέρη, ούτε το Ισραήλ, ούτε λόγω ανακοχή, γιατί νομίζω ότι έχουμε ανακοχή τώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να δεχτούμε ε, να σταματήσει η πρόταση ακριβώς όπως έχει ε, κατατεθεί τώρα. Σας ευχαριστούμε κύριε Ρωμανιούλη. Δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Γερζεμπόφσκι. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνεί η με την απόψη του κύριου Ρωμανιόλη. Είναι σημαντική αυτή η συμφωνία και για τις δύο πλευρές, όχι μόνο για το Ισραήλ και για την Παλαιστίνη, αλλά και για την δική μας οικονομία, για το δικό μας τουρισμό, για το δικό μας εμπορικό κόσμο και για το περιβάλλον. Χρειαζόμαστε στον τομέα της αεροπορίας ε, σωστές ρυθμίσεις και γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να προχωρήσουμε γρήγορα. Ήδη έχουμε καθυστερήσει. Νομίζω λοιπόν ότι καθοριστικό θα είναι όντω να υποστηρίξουμε και να υπερψηφίσουμε τη συμφωνία αυτή. Να σημειώσω κατά δεύτερον ότι η ομάδα μου απορρίπτει την ε, τροπολογία του κυρίου Τούσα γιατί ξεκινάει από λάθος ε, σημείο εκκίνησης. Θεωρεί ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση ξεκίνησε τις μάχες στη Γάζα. Θυμάμαι ότι η Χαμάς ε, εκτόξευε από το Λίβανο πυράβλους ε, στη Λωρίδα της Γάζας. Θα το έχει ξεχάσει ίσως ο κύριος Τούσας. Το θέμα της Μέσης Ανατολής, το θέμα της Λωρίδας της Γάζας δεν χρειάζεται να εισαχθεί εδώ στο θέμα αυτό. Το έχει τοποθετηθεί σωστά και ισορροπημένα το Κοινοβούλιο, με μεγάλη πλειοψηφία. Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν, άσχετα από το πώς βλέπουμε την σύγκριση, τη σύγκρουση αυτή, να αναχαιτήσουμε τη σημαντική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ. Γιατί και για τον αραβικό κόσμο είναι σημαντικό να προχωρήσουμε με τη συμφωνία αυτή. Γι' αυτό λοιπόν η δική μου ομάδα υποστηρίζει την έκθεση Ρωμανιόλη όσο έχει στην αρχή και γι' αυτό απορρίπτουμε την τροπολογία αυτή. Μάλιστα, ο κύριος Σίμψον. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Μιλώ εξ ονόματος του σκιώδους εισηγητή, ο οποίος δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μας εδώ. Εμείς μπορούμε να συμφωνήσουμε με την γραμμή την οποία προτείνει ο κύριος Ρωμανιόλη και μετά όσα είπε βέβαια ο κύριος Ζαρζεμπόφσκι τώρα. Οι δύο τροπολογίες που έχουμε εδώ πέρα πιστεύω ότι δεν σχετίζονται καν με τη συγκεκριμένη έκθεση αν η έκθεση αυτή είχε ως ζήτημά της την πολιτική κατάσταση στην Μέση Ανατολή και τις πρόσφατες εξελίξεις, τότε καταλαβαίνω ότι ναι, οι τροπολογίες αυτές μπορεί να ήταν και σχετικές. Αλλά εδώ μιλάμε για τη δημιουργία ενός κοινού αεροπορικού χώρου με το Ισραήλ. Επομένως, όσον αφορά τουλάχιστον την τροπολογία 1, θεωρούμε ότι δεν έχει θέση στην έκθεση αυτή, επομένως δεν μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Τώρα, όσον αφορά την τροπολογία υπαριθμών 2, όπου καλείται το Συμβούλιο και η Επιτροπή να διακόψουν άμεσα και να στείλουν διαπραγματεύσει με το Ισραήλ για τη σύναψη αυτής συμφωνίας. Εμείς ε, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε βέβαια κάτι τέτοιο στα πλαίσια της Επιτροπής μας, γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι θα εγκριθεί από την Επιτροπή μας αυτή η συμφωνία και συνέχεια ότι θα περάσει και στην Ολομέλεια. Τώρα, αν συμβεί κάτι στον ενδιάμεσο χρόνο στις σχέσεις μας με το Ισραήλ, και γενικότερα όσον αφορά την Μέση Ανατολή, τότε ε, ενδεχομένως να εξετάσουμε μία κάποια εναλλακτική λύση τότε όμως μόνο. Δηλαδή να πούμε ότι κοιτάξτε, δεδομένων των τελευταίων αυτών εξελίξεων δεν θέλουμε να υποστηρίξουμε τη σύναψη αυτής συμφωνίας με το Ισραήλ. Το βασικό όμω μήνυμα το οποίο πρέπει να προωθήσουμε είναι ότι τουλάχιστον όσον αφορά την διάσταση των μεταφορών θέλουμε να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με το Ισραήλ και γι' αυτό το λόγο υποστηρίζουμε τις προτάσεις του κ. Ρωμανιόλη. Τώρα, αν υπάρχουν ε, οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να προσθεθούν στην έκθεση αυτή, τότε νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να γίνει στην Ολομέλεια, όχι όμως τώρα στα πλαίσια της Επιτροπής των Μεταφορών, γιατί εμείς ως Επιτροπή των Μεταφορών πρέπει να αποφανθούμε για θέματα που αφορούν τις μεταφορές και για τίποτα άλλο κατά την άποψή μου. Τώρα, όσον αφορά την ε, πολιτική κατάσταση μέσα στην Ανατολή και όσον αφορά στα συμβάντα στην Γάζα, αυτά αποτελούν ξεχωριστό ζήτημα. Εμείς ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει στην έκθεση αυτή που αφορά τις μεταφορές να δώσουμε μία απάντηση, μία αντίδραση, η οποία θα είναι σχετική με το ζήτημα των μεταφορών. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Σας ευχαριστούμε πολύ. Δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Κράμερ. Ναι, η δική μου ομάδα στηρίζει επίσης την έκθεση του εισηγητή. Τα πολιτικά ζητήματα φυσικά είναι σημαντικά, αλλά δεν είμαστε πολιτική επιτροπή και δεν μπορώ καν να το διαβάζω το πόσο μονόπλευρα είναι εδώ πέρα οι τροπολογίες παρουσιασμένες. Δυστυχώς δεν είναι εδώ πέρα οι εισηγητές της τροπολογίας αν ήταν εδώ, θα ήθελα να τον ρωτήσω. Είναι υπέρ ή κατά του μομαρτισμού του Ισραήλ. Είναι υπέρ ή κατά της ανατείναξης των τούνελ. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα συζήτηση. Είναι μονόπλευρο. Μονόπλευρο και με ενοχλεί. Με ενοχλεί γιατί είναι δύσκολη η στιγμή που περάσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχαμε ένα ψήφισμα για την Παλαιστίνη και το Ισραήλ και ο πρόεδρος είχε στηρίξει με την ομάδα του το ψήφισμα. Έγινε κοινή δήλωση από όλες τις ομάδες. Έγινε ψηφοφορία χωρίς ούτε μία ψήφο κατά. Και ο πρόεδρος Πέτερινγκ, ο οποίος είναι εδώ από το 79, είπε ότι ποτέ ξανά δεν έχει δει παρόμοια κατάσταση. Και σε αυτή τη σύγκρουση λοιπόν, νομίζω ότι ως μικρή επιτροπή που δεν ασχολούμαστε με πολιτικά θέματα, δεν θα πρέπει να αναιρέσουμε το ψήφισμα αυτού του Κοινοβουλίου. και να αναφέρουμε ότι δεν θέλουμε περαιτέρω συμφωνίε με το Ισραήλ. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει στο σημείο αυτό να λάβουμε υπόψη την πολιτική άποψη του Κοινοβουλίου και να συμφωνήσουμε με την πρόταση του εισηγητή. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχει ζητήσει κανείς άλλο το λόγο. Συνεπώς, θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να καθυστερήσω άλλο. Α, συγγνώμη, Κομισιόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομο τόσο ή να σας πω απλώς ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, είναι σύμφωνη με όλες τις παρεμβάσεις που γίνανε σήμερα, σύμφωνη απόλυτα επίσης και με τον εισηγητή και όντως θεωρεί ότι ε, η έκθεση αυτή ασχολείται μόνο με την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη δημιουργία ενός κοινού αεροπορικού χώρου με το Ισραήλ και ότι προφανώς ε, οι διαπραγματεύσεις αυτές θα μπορούν να αφορούν και γενικότερα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να ληφθούν και τα οποία θα μπορούσαν να προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά στη φάση αυτή αυτό που μας ε, απασχολεί περισσότερο είναι η έναρξη των διαπραγματεύσεων αυτών, προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα κοινό αεροπορικό χώρο με το Ισραήλ. Επομένω, ε, υποστηρίζουμε τα όσα υπόθηκαν και προσβλέπουμε στη συνέχεια των ε, διαπραγματεύσεων. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα ναι κύριε Ρωμανιόλη έχετε όντω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να επαναλάβω λοιπόν τις ευχαριστίες στους συναδέλφους ε, και στον συνάδελφο Λιμπεράτσκι που με βοήθησε ως και ο τη γραμματεία και όλους εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Eh, e Ευχαριστούμε πολύ. Ας περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που έχει να κάνει με την απαλλαγή 2007 για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε και την απαλλαγή 2007 για τον Οργανισμό Ασφάλειας Αεροπορίας και τον Οργανισμό των Σιδηροδρόμων. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Κράμερ, ο οποίος είναι εισηγητής και για τα τρία αυτά σημεία. Νομίζω ότι μπορούμε και τις τρεις εκθέσεις να τις συζητήσουμε από κοινού, άλλωστε εκτενέστατα τις συζητήσαμε και σε προηγούμενες συνεδριάσεις μας. Δόθηκαν τότε πολλές διευκρινήσεις και είχαμε συμφωνήσει για τον τρόπο με τον οποίο θα εξετάζαμε τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Ορισμένες τροπολογίες έχουν ήδη εξεταστεί, Έχουμε και κάποιες νέες αυτή τη στιγμή. Γνωρίζουμε ποια είναι τα προβλήματα που έχουν οι οργανισμοί αυτοί. Προτείνουμε να δοθεί απαλλαγή και στους τρεις οργανισμούς, λέγοντας όμως ότι προσβλέπουμε σε καλύτερη διαχείριση των ταμείων και γενικότερα των πόρων στο μέλλον. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τους και Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει ο κ. Γερζεμπόφσκι εξ του ΕΛΚ. Μάλιστα, πολύ ωραία. Τι ωραία που συμφωνούμε όλοι μαζί. Τουλάχιστον ε, θα ήταν πολύ ωραία να καταφέρουμε να συμφωνούσαμε. Μπορούμε να δεχθούμε την ε, τροπολογία Γιάνσεν. Όσον αφορά τώρα την τροπολογία 2, νομίζω ότι ε, εδώ πέρα η έκθεση είναι αρκετά αυστηρή, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει λοιπόν τροπολογία αυτή. Όσον αφορά τις τροπολογίες των φιλελευθέρων, νομίζω ότι έχουν ένα πολύ ακαδημαϊκό δασκαλίστικο χαρακτήρα. Μοιάζει να απευθυνόμαστε στους οργανισμούς αυτούς λέγοντας ότι εμείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασκήσει πίεση στους οργανισμούς αυτούς προκειμένου να διατελέσουν σωστά την εργασία τους. Νομίζω ότι η έκθεση του κυρίου Κράμερ μιλάει από μόνη της και πολλές φορές διαφοροποιεί τον έναν οργανισμό από τον άλλον. Σαφώς θα μπορούσαμε να προσάψουμε διάφορα πράγματα στους οργανισμούς αυτούς, ότι δεν καταφέραν να διαχειριστούν πολύ καλά τον προπολογισμό τους και διάφορα άλλα πράγματα. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε από κοινού και τόσο απλουστευτικά να κατηγορούμε και τους τρεις οργανισμούς μαζί. Ξέρετε ότι στο παρελθόν πολλές φορές τα προβλήματα των οργανισμών αυτών είχαν να κάνουν, όπως το είπε και η κυρία Γιάνσεν, με το ότι ε, οι οργανισμοί αυτοί δεν κατάφερναν να επιλέξουν καλά το προσωπικό τους. Και αυτό γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε θέσει ένα λανθασμένο πλαίσιο επιλογής προσωπικού για αυτούς τους οργανισμούς. Όσον αφορά τον Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, θα ήθελα να σας πω ότι ναι, ενδεχομένως να διέπραξε κάποια λάθη ο οργανισμός αυτό στο παρελθόν, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αυτή, ήταν η μόνη υπεύθυνη για τη διόρθωση των λαθών αυτών. Θεωρώ πάντως ότι η τροπολογία αυτή είναι ιδιαίτερα υπερβολική και ο έντονος χαρακτήρας σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται. Άλλωστε, μιλάμε, συζητάμε εδώ πέρα για μια γνωμοδότηση η οποία απευθύνεται στην Επιτροπή Προπολογισμών επαναλαμβάνω πάντως ότι ε, η έκθεση Κράμερ είναι πολύ καλή και νομίζω ότι στοχεύει σε κάθε οργανισμό ξεχωριστά, εντοπίζοντας θετικά και αρνητικά σημεία για κάθε οργανισμό ξεχωριστά. Εμείς προτείνουμε γενική απαλλαγή λοιπόν και για τους τρεις οργανισμούς. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αποδεχθούμε το δασκαλίστικο τόνο των τροπολογιών των σοσιαλιστών. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο δίνω στον κύριο Σίμψον εξ ονόματος των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα η άποψη των χριστιανοδημοκρατών που πιστεύουν ότι δεν θα πρέπει να έχουμε αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία με τα λεφτά του φορολογούμενου πολίτη. Αυτό προκύπτει από τα όσα είπε ο κύριος Γαρζεμπόφσκι. Εγώ νόμιζα ότι οι φίλοι του στις τράπεζες μπορεί να έχουν άλλα πράγματα να μας πούνε, αλλά τέλος πάντων για το θέμα μας. Ο οποιοδήποτε ήταν παρόν σε αυτή τη συνεδρίαση και δεν ξέρω για οργανίσουν εδώ όταν ε, συζητούσαμε αυτούς τους οργανισμούς αυτό το οποίο κατέστη σαφές καταφανές ήταν ότι υπάρχει πρόβλημα και οι οργανισμοί δεν τηρούν τον προπολογισμό τους. Έχουν προβλήματα στην τηρήση του προπολογισμού τους, ε, ξεπερνούν τον προπολογισμό, ως προς το προσωπικό υπάρχουν πολλά προβλήματα, για προσωπικό το οποίο ε, προσλαμβάνεται ή δεν προσλαμβάνεται. Μια ανακατοσούρα πραγματικά. Εγώ δεν είμαι διατεθειμένος λοιπόν να κάτσω εδώ με τα λεφτά του Ευρωπαίου Φορολογούμενου και να λέω ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και δεν θα πρέπει να είμαστε πολύ ε, ελαστικοί με αυτούς τους ανθρώπους των ε, οργανισμών. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση ως ε, δημοσιονομική αρχή και ως αρχή ελέγχου του προπολογισμού να δεχτώ κάτι τέτοιο δεν επικρίνουμε κανέναν οργανισμό, δεν λέμε ότι θα πρέπει όλους να τους ε, κλείσουμε ή να τους ε, κάψουμε στην πυρά. Απλά και μόνο λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι ο οργανισμός θα πρέπει να διατηρήσει την αυστηρή δημοσιονομική του πειθαρχία στο μέλλον και να δουλεύει με βάση το συμπεφωνημένο προπολογισμό. Αν όλα αυτά σας φαίνονται βαριά, τότε θα έπρεπε να δείτε την αρχική διατύπωση. Τότε θα είχατε δει τι έγραφα. Αλλά αυτή είναι απλή μια απόπειρα να θέσω τις συζητήσεις που έγινα τότε όπου ήταν σαφές όχι μόνο για μένα και τη δική μου πλευρά αλλά και για όλους όσους ε, κάθονται εδώ στο, ε, στην αίθουσα ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη δημοσιονομική πειθαρχία και αν θέλετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μπορέσει να διατηρήσει αυτή τη δημοσιονομική πειθαρχία. Αυτά ε, επικύψαν και αυτέ είναι οι τροπολογίε. Όσον αφορά τώρα τι τροπολογίε τη κυρία Γένσεν, αυτέ νομίζω ότι προέκυψαν από την ε, δεύτερη, αν θέλετε, φάση αναταραχή που ήταν το θέμα του προσωπικού. Που και πάλι άφηνε πάρα πολλέ εκκρεμότητε και υπήρχε το εξή σενάριο. Να προσλαμβάνουμε κάποιου με μερική απασχόληση και μετά να μην του προσλαμβάνουμε, μετά να προσλαμβάνουμε κόσμο και μετά να έχουμε μια ολόκληρη έκθεση που μα λέει ότι υπάρχουν ελλείψει. Κατανοώ τα όσα λέει η κυρία Γένσεν λοιπόν. Ουσιαστικά το μόνο που θέλουμε να πούμε σε αυτούς τους οργανισμούς και να πούμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εμείς που σας, ε, ε, είμαστε πίσω από το λαιμό σας, πίσω από το σβέρκο σας και σας παρακολουθούμε για τον προϋπολογισμό θέλουμε να κάνετε τα όσα σας δίνονται, να χρησιμοποιείτε τα κονδύλια που σας δίνουν και να έχετε δημοσιονομική πειθαρχία. Αν θεωρείτε ότι είναι πολύ βαριά η διατύπωση, ναι, δηλώνω ένοχος, αλλά από εκεί και πέρα ελπίζω ότι η Επιτροπή θα μας υποστηρίξει. Και εκεί να δείτε τι θα γίνει με την Επιτροπή Πολυβολογισμού. Εκεί είμαι 100% βέβαιος ότι θα μας υποστηρίξουν. Ε, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γένσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Διάβασα την έκθεση του κυρίου Κράμερ. Θα συμφωνήσω με τις δικές μου τροπολογίες και τις τροπολογίες του κυρίου Σίμψον. Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο δύσκολες. Είναι προφανές νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει δημοσιονομική πειθαρχία στον τομέα αυτό. Αλλά θα πρέπει να σας πω ότι οι τροπολογίες μου προέκυψαν από τις συζητήσεις που κάναμε. Υπάρχουν προβλήματα με τους οργανισμούς αυτούς και πολύ συχνά μπλέκονται, αν θέλετε, μεταξύ των διάφορων φορέων. Έχουν τεράστια, τεράστιες επιτροπές από το Συμβούλιο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες και οι όροι. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να αποτυπώνεται και στις σχέσεις μας με τους οργανισμούς αυτούς. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπερψηφίσουμε τις δύο αυτές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη συζήτησή μας. Να δώσω το λόγο στον κύριο Μπονούτσι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μετά στον κύριο Κράμερ για να κλείσει τη συζήτηση. Thank uh, uh, uh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχω να σας πω ότι εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την ε, τροπολογία που προτείνει ο κύριος Σίμψον. Είναι αυτονόητο ότι είμαστε υπέρ της επέκτασης των τριών οργανισμών εντός του πλαισίου προϋπολογισμού που έχουμε θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουν το προσωπικό που τους χρειάζεται. Σαφώς πρέπει να υπάρχει πειθαρχία και αυτό είναι μονόδρομος. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε για τη διασφάλιση προσωπικού το 2006 και το 2007 έχει περάσει πλέον εισερχόμαστε σε μία φάση όπου μπορεί πλέον ο οργανισμός ε, να συνεχίσει τις ε, συνήθεις εργασίες του με σταθερό τρόπο και αυτό εντός ε, των προβλέψεων του προπολογισμού που έχουμε κάνει για τώρα, από τώρα μέχρι το 2013. Δυστυχώς υπήρξε μια μείωση πέρσι για όλους τους οργανισμούς κατά 50 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι χρειάστηκε να αναθεωρήσουμε τις δυνατότητες για όλους τους για τα επόμενα ε, χρόνια, αλλά μπορούμε κάλλιστα σε περίπτωση που το αποφασίσει η αρχή προπολογισμού να χρησιμοποιήσουμε το αποθεματικό ή να ανακατευθύνουμε κάποια από τα προγράμματα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή σε λειτουργία. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Ο Κράμερ. Ωραία λοιπόν να το παίξει ο σε ό,τι αφορά τις ερμηνείες που είπατε κύριε Γιαζεμπόφσκι τι λέμε ότι καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει ότι ο οργανισμός στο μέλλον θα εφαρμόσει αυστηρή δημοσιονομική επιθεραχία και εντός του πλαισίου το οποίο έχει συμφωνηθεί να εργαστεί. Αυτό δεν λέει παρά το αυτονόητο. Αυτό δηλώνει μόνο. Θα σας κάνω εγώ μάθημα τώρα. Να ερμηνεύσουμε εμείς λοιπόν. Τι να κάνω να πω στον μαθητή Γιατζεμπόφσκι ότι με τη δημοσιονομική αυτή πειθυρχία που αναφέρει κάθε νόμος να τα αφήσουμε και να κλείσουμε αν θέλετε και να γυρίσουμε την πλάτη σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτή είναι η πρότασή σας. Αυτό προτείνετε να κάνουμε. Όχι. Είμαι αυστηρός καθηγητής και με υποστηρίζει και ο καθηγητής ε, Σίμψον και η Δανέζα συνάδελφος. Είναι το προφανές. Μπορούμε να το γράψουμε, μπορούμε να το αφήσουμε, αλλά δεν επηρεάζεται καθόλου η κριτική με την πρόταση αυτή που, προσθέ, που προσέθεσα. Não quero deixar de manifestar a minha satisfação porque esta é uma comissão enriquecida. O número de pessoas. Ναι, είμαι πολύ ικανοποιημένο, λέει ο Πρόεδρο που έχουμε τόσο καλούς βουλευτές εδώ πέρα στην Επιτροπή μας που εμπλουτίζουν τη συζήτηση. Κρίσια Ζεμπόφσκι, κύριε Κράμερ, όταν κάνατε μία έκθεση το 2009 που υποδεικνύεται τα ελλείμματα δικαίως και υποστηρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρέπει να επαναλάβει τα ίδια σφάλματα. Όλα αυτά καλά και ωραία. Όταν λέμε όμως στο τέλος ότι το 2009, για μια έκθεση του 2007, έτσι, ότι καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον, το οργανισμός να εφαρμόσει αυτή τη δημοσιονομική επιτυχία. Τι σημαίνει δηλαδή ότι το 2007, 2008 και 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο οργανισμός δεν ακολούθησε την αυστηρή δημοσιονομική επιταρχία που έπρεπε. Δεν μπορούμε να αποφθύνουμε τέτοιες κατηγορίες γιατί το θέμα είναι το κατά πόσον αρκεί να κάνουμε κριτική στους ε, οργανισμούς αυτούς και μετά ερχόμαστε και σαν καθηγητές να λέμε ότι κοιτάξτε πειθαρχία και εσύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στραβάμε τα αυτή. Εγώ σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα αντιδρούσα έτσι. Εγώ τι θα έλεγα, ότι εμείς φροντίζουμε πάντα οι οργανισμοί να εργάζονται με τη Μοσονομική επιθαρχία και δεν χρειαζόμαστε επιπλέον ε, εκκλήσεις, αλλά ευτυχώς είναι λίγο πιο ευγενική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν παρεκτράπηκε και η συζήτηση. Ο λόγος του κύριο Σίμψον για να ολοκληρώσει τη συζήτηση. Κύριε Πρόεδρε, είναι φρικτή η σκέψη να συμφωνήσει ο Γιώργη με την Κομισιόν. Θα σταματήσω τώρα. Δε, θεωρώ ότι δεν συνέβη ποτέ αυτό, διότι αλλιώς όλη η διαδικασία θα κινδυνεύει. Θα τηρήσουμε την τροπολογία μας. Ευχαριστώ. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Η οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών. Να δώσω το λόγο στο συντάκτη της γνωμοδότησης, τον κύριο Μπλόκλαντ. Κύριε Μπλόκλαντ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αύριο θα ψηφίσουμε για τη γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Απασχόλησης για την ε, οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελέντων κινητέ δραστηριότητε οδικών μεταφορών. Και θα είναι πολύ βασική η ψηφοφορία αυτή, γιατί θα συμπεριληφθούν οι αυτοαπασχολούμενοι ή όχι. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι οι πραγματικοί αυτοαπασχολούμενοι θα πρέπει να παραμείνουν εκτός του πεδίου εφαρμογή της οδηγίας. Πέρα από το γεγονός ότι ο χρόνος εργασίας ε, των αυτοαπασχολούμενων δεν μπορεί να παρακολουθηθεί, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν θα συμβάλλει καθόλου στην οδική ασφάλεια τελικά μια τέτοια ρυθμίση για την οδική ασφάλεια. Χρειαζόμαστε, μάλλον υπάρχει ήδη ε, ε, για την ασφάλεια και την, τους σε ό,τι αφορά τον χρόνο εργασίας. Αυτό συμβάλλει στην ασφάλεια, στην οδική. Και η συμπερίληψη των αυτοπασχολούμενων δεν θα συμβάλλει στην οδική ασφάλεια ας προσπαθήσουμε να καταρτήσουμε μία οδηγία η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα μια καλή σχέση μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου. Να είναι σαφής η νομοθεσία, με σαφείς ορισμούς, σαφείς ρυθμίσεις, περισσότερη συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών για την πρόληψη των, του φαινομένου των ψευδοπασχολούμενων. Όταν, ε, λάβουμε υπόψη τα θέματα αυτά, θα προωθήσουμε την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων και θα συμβάλλουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς. Σας είπα στην αρχή ότι θα είναι σημαντική η ψηφοφορία αύριο, γι' αυτό δεν υπέβαλα και συμβιβαστικέ προτάσεις. Δεν είναι εύκολη η εξέβρεση συμβιβασμών για το κατά πόσο θα συμπεριληφθούν οι μη οι αυτοπασχολούμενοι για την συνάδελφό σου Γκερέιρερ, Κουστάτσερ, του ΣΑΣ κτλ. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με τις τροπολογίες σας, γιατί θεωρώ ότι οι τροπολογίες αυτές δεν συμβάλλουν ε, στη διαμόρφωση ξεκάθαρων όρων και θεωρώ ότι και η επιχειρηματολογία σας δεν είναι αρκετά πιστική. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία υπαριθμών 12, γίνεται αναφορά κεφάλαιο 3.2 του 2007-266 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναφέρεται λοιπόν το εξής. Οι σύμβουλοι υποδεικνύουν ότι η οδική ασφάλεια μπορεί να ωφεληθεί πιο πολύ αν συμπεριληφθούν άλλοι παράγοντες, όπως για παράδειγμα καλύτερη τήρηση του χρόνου ε, οδήγησης, παρά σε ό,τι αφορά τη μείωση του χρόνου εργασία για τους αυτοπασχολούμενους οδηγούς. Τέλος παράθεσης. Επίσης, να σας αναφέρω τι λέει η έκθεση, το κεφάλαιο 3.5 της έκθεσης αυτής. Δυστυχώς λοιπόν δεν με πείθουν τα επιχειρήματα του συναδέλφου σε ό,τι αφορά τον ορισμό της νύχτας. Ίσως να ήταν δυνατή η εξέβρεση συμβιβασμού, αλλά όλες ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η έκθεσή μου και οι τροπολογίες ε, των συναδέλφων ορίζουν τη νύχτα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει μεταξύ ε, μεσάνυχτα και 7 το πρωί με μίνιμουμ 4 ωρών. Έχουμε τους αδελφούς Κούστατσερ και Γκερέρο, οι οποίοι προτιμούν πιο μακριές νύχτες από τις 10 η ώρα το, το βράδυ μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί ή και από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 7 το πρωί. Στην τροπολογία μου υπαριθμών 3 ε, ακολούθησα τη μέση οδό. Μία νύχτα μεταξύ 12 και 7 μεταξύ 12 και 6, η οποία αποτελείται τη χρυσή τομία, αν θέλετε. Και θεωρώ ότι έτσι δευκρινίζεται και ο όρος της νύχτας σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί. Να καλέσω τους συναδέλφους, λοιπόν, να υπερψηφίσουν την τροπολογία μου υπαριθμών 3 θεωρώ ότι αυτό και ευελιξία επιτρέπει και διαφάνεια σε ό,τι αφορά το περιθώριο των τριών ωρών για την νυχτερινή εργασία θα πρέπει να διατηρηθεί γιατί ένας οδηγός ο οποίος έχει δουλέψει όλη την ημέρα και λόγω ανώτερης βίας αναγκάζεται να δουλέψει λίγο παραπάνω δεν πρέπει να αντιμετωπίζει κατευθείαν ε, το μειονεκτικό καθεστώς, αν θέλετε, της νυχτερινής εργασίας. Η νυχτερινή εργασία έχει προβλεφθεί για να προστατεύει τους εργαζόμενους από την εργασία κατά τη διάρκεια της νύχτας, όχι για να τους δημιουργεί προβλήματα αν υπάρχει κάποια, κάποιο απρόβλεπτο γεγονός. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει να εγκρίνουμε τις ε, τροπολογίες 34-35 σε ό,τι αφορά την ε, σωστή υποπτία της οδηγίας αυτής. Είναι σημαντικό τμήμα της οδηγίας και να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Γιάκοψη για την τροπολογία περιθμών 40 που υποβολή, υπέβαλε. Ωστόσο, πολύ φοβάμαι ότι θα προκύψουν ε, γραφειοκρατικά άχθη για τις ε, εθνικές ε, διοικήσεις. Νομίζω ότι καλύτερη είναι η πρόληψη από ότι η εκ των υστέρων αντιμετώπιση, αλλά νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Ξέρουμε λοιπόν ποια είναι στο ευρωπαϊκό επίπεδο η λύση. Να κοιτάξουμε τον, την οδηγία για το χρόνο εργασίας. Αυτή να προωθήσουμε, αυτή να εφαρμόσουμε και μετά αυτή την οδηγία. Έτσι θα καταστούν πιο ασφαλείς οι ευρωπαϊκές οδοί και θα δημιουργηθεί μια καλή σχέση μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη στον τομέα αυτών. Τέλος, τρεις ε, παρατηρήσεις ε, επιτρέψτε μου. Η τροπολογία 16 του κυρίου Κουστατσέρ, πολύ καλή τροπολογία, αλλά αναφέρεται ήδη στο άρθρο 11 της ε, οδηγίας αυτής ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι αποτρεπτικά και αναλογικά. Νομίζω ότι αυτό επαρκεί. Και κατά δεύτερον θα σημειώσω επίσης ότι έχω αποσύρει την τροπολογία 2 γιατί θεωρώ ότι δεν συμβαδίζει με άλλες ρυθμίσεις ό,τι αφορά τον χρόνο εργασίας. Χαίρομαι που την προηγούμενη φορά συζητήσαμε το σημαντικό αυτό θέμα, γιατί ως απόρρια της συζήτησης α, αυτής θεωρώ ότι προέκυψε η τροπολογία υπερθμών 31 της ε, κυρίας Παναγιωτοπούλου που θα υποστηρίξετε τους υποεργαζόμενους και τους εργοδότες αυτούς που εμπλέκονται στα θέματα αυτά. Και τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Γραμματεία για την εξαιρετική συνεργασία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Eh, Ευχαριστούμε πολύ και δίνω το λόγο immer leicht, deshalb möchte Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να αναφερθώ στο σύνολο της έκθεσης βάσει κάποιων τροπολογιών που έχουν υποβληθεί. Αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας είναι μία πρόταση η οποία επηρεάζει όλους αυτούς που πειράζονται και από τους κανόνες για το χρόνο ανάπαυσης. Αν για παράδειγμα οδηγείτε φορτηγό το οποίο είναι άνω από ένα επίπεδο 3,5 τόνου θα πρέπει να συμμορφώνεστε με συγκεκριμένους κανόνες. Με διαφορετικούς κανόνες θα πρέπει να συμμορφώνεστε αν το φορτηγό το οποίο οδηγείτε είναι από 4,5 τόνους και πάνω. Πάντα αναφερόμενο στον χρόνο άπαυσης. Αν δούμε το άρθρο 16 του 93 104 βλέπετε ότι Πολλά από τα όσα προβλέπονται στην έκθεση αυτή αποκλείονται. Τέσσερι τροπολογίε έχω αποβάλει εγώ για να καταστεί το κείμενο πιο συγκεκριμένο. Πρώτον, η εργασία κατά τη διάρκεια τη νύχτα, τα όσα προβλέπονται τουλάχιστον για την εργασία αυτή, δεν θα πρέπει να τροποποιηθούν, δηλαδή να διατηρήσουμε τη χρονική διάρκεια από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 7 το πρωί και το ίδιο να ισχύει και για την εργασία κατά τη διάρκεια τη εβδομάδα. Κατά δεύτερον, χρειαζόμαστε σαφή διάκριση μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη και νομίζω ότι το θέμα των ψευδαπασχολούμενων αποτελεί αρμοδιότητα των εθνικών κρατών μελών. Αυτοί θα πρέπει να εξετάζουν κατά πόσον υπάρχουν ή όχι οι ψευδαπασχολούμενοι. Γι' αυτό θεωρώ ότι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σημείο αυτό είχε υποβάλει σαφή πρόταση όπως έγινε και στο άρθρο 2 στην οδηγία του Μαρτίου του 2004 θα έπρεπε να πει ότι θεωρούμε ότι οι αυτοαπασχολούμενοι εξαιρούνται τελεία και παύλα. Το τρίτο που θα προτείνω ωστόσο είναι το εξής. Δεν έχει συζητηθεί τόσο πολύ. Ποιος χρόνος εργασίας ισχύει για το προσωπικό σε ό,τι αφορά τις οδικές μεταφορές στο 3,5, σε ό,τι αφορά τους μισθωτούς δηλαδή. Στο σημείο λοιπόν αυτό θα μπορούσαμε να επιλύσουμε το κενό που υπάρχει λέγοντας ότι η οδηγία για το χρόνο εργασία αφορά κάθε εργαζόμενο ο οποίος ε, εμπλέκεται στην οδική, στις οδικές μεταφοράς που υπάρχει στο 3,5 και σε ό,τι αφορά το 3,8 συγγνώμη και τους ε, αυτοαπασχολούμενους ε, τους καλύπτει το 3,5. Αυτό θα ήταν σαφές και στην περίπτωση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να ορίσει κατά πόσο ο χρόνος ανάπαυσης ε, καθορίζεται από το 3,8 γιατί ήταν και πολύ οριακή ψηφοφορία εδώ στο Κοινοβούλιο από ό,τι άκουσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γίνονται σχετικές μελέτες και έρευνες. Αν η ασφάλεια αλλάξει το όριο των 3,5 τόνων. Αυτό λοιπόν δεν θα επηρεάσει την οδηγία αυτή. Αυτό θα επηρεάσει κάποιους άλλους ε, οδηγούς, τους οδηγούς εξπρέ, όπως ε, αναφέρονταν, αλλά δεν θα επηρεάσει τους χρόνους αναπαυσής. Αυτό όμως αποτελεί κάτι μεροντικό. Θα ήθελα λοιπόν να πω το εξή. Οι προτάσεις μας θέλουν να προσθέσουν σαφήνεια οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν συμπεριλαμβάνουν τα αυτονόητα. Το ΕΛΚ δεν ε, έχει πρόβλημα, αλλά καλό θα ήταν να υπήρχε μια οδηγία για το χρόνο εργασία για όλους ε, τους απασχολούμενους και σε ό,τι αφορά το όριο των 3,5 τόνων. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί κάτι το προφανές για όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Γιάκοψ. Κυρία Γιάκοψ, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής είχαμε εξετάσει τις προτάσεις και ευχαριστούμε τον κύριο Μπλόκλαν για τις εξηγήσεις που μας έδωσε γιατί εξήγησε και παρουσίασε για μια ακόμη φορά τα αμφιλεγόμενα σημεία Θεωρώ και θεωρούσαν δηλαδή και από πριν ότι σημαντικά ήταν κάποια ζητήματα σε ό,τι αφορά του κατά πόσο θα συμπεριληφθούν στην οδηγία οι αυτοαπασχολούμενοι. Ο κ. Μπλόκλαντ ανέφερε ότι πρόκειται για ένα θέμα επί της αρχής. Σας είχα πει ότι θα διαβουλευτούμε και με τους κοινωνικούς εταίρους, το οποίο και πράξαμε διεξοδικά. Κατέληξα λοιπόν στο συμπέρασμα ότι θα ήταν πραγματικά ανεύθυνο να μην συμπεριληφθούν οι αυτοπασχολούμενοι στην οδηγία αυτή και θα ήθελα να το διευκρινίσω αυτό και να το αναλύσω. Αν δεν συμπεριληφθούν οι αυτοπασχολούμενοι στην οδηγία αυτή, υπάρχονται ουσιαστικά μόνο στην ε, οδηγία για το χρόνο ανάπαυση. Πολλοί θεωρούν ότι αυτό αρκεί, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες μου αυτό θα καθιστούσε δυνατόν Ε, η εργασία να ξεπεράσει να προσθεθεί εργασία 84% και πάνω. Και όχι μόνο σε ό,τι αφορά ε, τις οδικές μεταφοράς, αλλά και διοικητικά θέματα. Και σε οποιασδήποτε άλλες περιπτώσεις θα ήμουν λιγότερο διαλλακτική, θα ήμουν περισσότερο διαλλακτική. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για την οδική ασφάλεια. Δεν είναι δυνατόν να είναι εξαντλισμένη η οδηγή των φορτηγών μετά από τεράστιες εβδομάδες, τεράστιες ημέρες και να προκαλούν θαντιφόρα ατυχήματα. Η οδική ασφάλεια αποτελεί ένα γενικό κοινωνικό θέμα και αυτό υπερέχει του οικονομικού συμφέροντας του αυτοαπασχολούμενη στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί σε ορισμένε περιπτώσει θα πρέπει να προστατεύουμε τον άνθρωπο από τον ίδιο του τον εαυτό. Πώ να το κάνουμε. Και επίση το γνωρίζουμε αυτό, γι' αυτό έχουμε προβλέψει άλλωστε και τον χρόνο ανάπαυση κτλ. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε υπέρ της συμπερίληψης των αυτοπασχολούμενων στην οδηγία αυτή. Υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία για τα οποία υπέβαλα τροπολογία σε ό,τι αφορά τον, ε, τη νύχτα. Προσπαθώ να κάνω λίγο πιο συγκεκριμένη την πρόταση του κυρίου Μπλόκλαντ. Επίσης το θέμα της εποπτείας είναι πολύ σημαντικά γιατί όλοι συμφωνούμε ότι δεν επαρκεί η φυστάμενη εποπτεία. Και τέλος, αν δεν ε, καταφέρουμε να συμπεριλάβουμε τους αυτοπασχολούμενους στην οδηγία, οι σοσιαλιστές προτιμούν την υφιστάμενη οδηγία για τους αυτοπασχολούμενους, για την αυτόματη υπαγωγή τους στο πεδίο της οδηγίας αυτής, γιατί ορίζεται άλλωστε και από την πολιτική και θα τεθεί σε εφαρμογή από το Μάρτιο. Ευχαριστούμε. Κυρία Γιάνσεν από την ομάδα Άλντε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι η δική μου πολιτική ομάδα συμφωνεί περισσότερο με τον κύριο Γκόσπ από ότι με την κυρία Γιάκοψεν για το ζήτημα αυτό. Τώρα, αν θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι αυτοπασχολούμενοι, Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο να το ελέγξει κανείς, δηλαδή να ελέγξει κανείς την εβδομάδα εργασία των αυτοπασχολούμενων, όπως και για μας. Καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές οι αυτοπασχολούμενοι χρησιμοποιούν τον ελεύθερό τους χρόνο προκειμένου να καθορίσουν ε, τα λογιστικά του στοιχεία. Είναι πολύ δύσκολο να καταφέρει, για να, να, καταφέρει να κρίνει κανείς για ένα αυτοπασχολούμενο τι είναι πραγματικός χρόνος εργασίας και τι όχι. μπορούμε να υποστηρίξουμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τους, λε, τους λεγόμενους για του οδηγούς φορτηγών συγκεκριμένα βέβαια και σαφώς είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανείς σωστή διάκριση, είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανείς σωστό έλεγχο. Θεωρούμε λοιπόν ότι μέσω τροπολογία θα πρέπει να λέμε ότι ε, προκειμένου να τηρήσει κανείς τους κανόνες για τους αυταπασχολούμενους θα πρέπει να λάβει υπόψη και την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία. Πέραν τούτων, θεωρώ ότι θα πρέπει να τηρηθούν οι υφιστάμενοι κανόνες όσον αφορά την εργασία κατά τη διάρκεια της νύχτας, ότι δεν θα πρέπει να τροποποιήσουμε τίποτα όσον αφορά την Κυριακή. Και ουσιαστικά πιστεύω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τις τροπολογίες και τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής με κάποιες διευκρινήσεις βέβαια Βέβαια, βλέποντας πώς εξελίσσει η συζήτηση στην Επιτροπή Απασχόλησης, θεωρώ ότι θα είναι δύσκολο να καταφέρουμε να διατηρήσουμε το υφιστάμενο κείμενο και τις προτάσεις σας. Φοβάμαι ότι ε, πάρα πολλοί τελικά δεν γνωρίζουν ότι ε, καλύπτονται από τις οδηγίες για το χρόνο ανάπαυσης και την οδηγία για το χρόνο εργασίας. Πάντως, ε, ο κατάλογος ψηφοριών που θα προτείνουμε θα αντικατοπτρίζει και τις θέσεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση στο σημείο αυτό, δίνω το λόγο στον κύριο Στάτσεκ, στο των Πρασίνων. Ευχαριστώ κύριε Κούστατσερ. Οι πράσινοι προσεγγίζουν μάλλον τους σοσιαλδημοκράτες παρακολούθησα και τη συζήτηση στην Επιτροπή Απασχόλησης κινείται μάλλον προς την κατεύθυνση να απομακρυνθούμε ακόμα πιο πολύ από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να επισκνάσουμε την πρόταση αυτή μετά από ποιήση του Συμβουλίου. Αλλά πιστεύω ότι αν θα πρέπει, αν λαμβάνουμε στα σοβαρά την ανθρώπινη ζωή και τα ατυχήματα που γίνονται στο δρόμο, και κυρίως τα ατυχήματα που προκαλούνται και από τα μεγάλα φορτηγά θα πρέπει πραγματικά να τα λάβουμε αυτά σε σοβαρά και να είναι πιο σοβαρές και αυστηρές ρυθμίσεις μας. Αν θέλουμε να ελέγξουμε τους πασχολούμενους, μπορούμε να ελέγξουμε και τους αυτοπασχολούμενους. Αυτό είναι σαφές, αλλά Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, η ανάπαυση κατά τη νύχτα, το, κατά το Σαββατοκύριακο, θα πρέπει να τηρούνται. Αν λέμε δηλαδή ευθύ εξ αρχή ότι αυτό δεν μας ενδιαφέρει, δεν θέλουμε να το ελέγξουμε, ξέρουμε ότι θα χαλαρώσει κι άλλο η κατάσταση στην Επιτροπή Απασχόλησης ακούγονται κάποια στοιχεία που διασαφηνίζουν, μάλλον που αποδυναμώνουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ θα ήθελα να είμαστε πιο αυστηροί και να παρακολουθήσουμε και να θεωρήσουμε το όλο θέμα υπό το πρίσμα της οδικής ασφάλειας. Όχι πώς θα βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις, όχι πώς θα βοηθήσουμε τα συνδικάτα, αλλά με απότερο σκοπό την οδική ασφάλεια. Είμαι πεπισμένος λοιπόν ότι χρειαζόμαστε πιο αυστηρούς κανονισμούς, όχι πιο χαλαρούς κανονισμούς. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, νομίζω ότι μίλησαν όλοι που ήθελαν να πάρουν το λόγο. Θα ακούσουμε τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Μπλόκλαντ, το συντάκτη μάλλον, για μια γνωμοδότηση την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί πάρα πολύ χρήσιμη και παρουσιάστηκαν και κάποιε τροπολογίε που μπορεί να υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι θεωρεί ότι ενισχύουν τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα προκειμένου να δώσουμε σε εφαρμογή καταλήλω την νομοθεσία. Καταρχάς να σας υπενθυμίσω ότι όταν η πρόταση της οδηγίας 2008-0195 ε, προτάθηκε το 1998, οι αυτοαποσχολούμενοι οδηγοί ε, είχαν προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένας τρόπος για να ενισχύσουμε αυτό που θεωρούσαμε ανεπαρκές, ακατάλληλο, μη ικανοποιητικό εφαρμοστικό πλαίσιο των όρων, των ορών οδήγησης και των χρόνων ξεκούρασης που ίσχυαν τότε. Τώρα η κατάσταση έχει αλλάξει σημαντικά. Έχουμε μια νέα στεναρή νομοθεσία για τις ε, ώρες οδήγησης και τους χρόνους ξεκούρασης, ε, μια, ένα κανονισμό ο οποίος εγκρίθηκε πριν από κάποια χρόνια, ο οποίος Ισχύει για όλους τους οδηγούς. Είτε είναι υπάλληλοι είτε είναι αυτοαποσχολούμενοι. Η οδήγηση και η φροντίδα του ε, φορτηγού οχήματος αποτελεί ε, τουλάχιστον ε, το μισό χρόνο των οδηγών είτε είναι αυτοαποσχολούμενοι είτε είναι υπάλληλοι. Ούτως ή άλλως λοιπόν το τμήμα της οδήγησης ε, καλύπτεται και από τις ώρες οδήγησης ε, των, ε, των καλύπτεται και για τους υπαλλήλους. Έχουμε επίσης ένα κανονισμό ο οποίος έχει πιο αυστηρά πλαίσια από την προϋπάρχουσα νομοθεσία. Θεωρούμε λοιπόν ότι και εδώ έχουμε προχωρήσει. Επίσης η εισήχθη ο ψηφιακός ταχογράφος. Ε, φαίνεται ότι μπορεί να δημιουργεί και κάποια προβλήματα διότι είναι υπερβολικά ακριβής κατά την ε, καταγραφή του χρόνου οδήγησης για τους ε, οδηγούς. Νομίζω λοιπόν ότι η κατάσταση έχει αλλάξει εκ βάθρων και θεωρούμε ότι πλέον υπάρχουν εγγύησει προκειμένου να μπορέσουμε να περάσουμε στο γενικό κανόνα. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το θέμα μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ως προς τον γενικό κανόνα για το χρόνο εργασίας η οδηγία για το γενικό χρόνο εργασίας αποκλείει τους αυτοαποσχολούμενους. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα από όσα προβλέπει η γενική οδηγία για το χρόνο οδήγησης. Έγινε μία μελέτη, κάναμε αρκετές μελέτες, συμμετείχαν ενδιαφερόμενοι Ίσως να μην έγινε επίσημη, αλλά έγινε μια μακροσκελέστατη άτυπη συζήτηση με τους ενδιαφερομένους και αυτό το οποίο κατέστησε σαφέ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι δεν πρόκειται να αποκομίσουμε κανένα όφελος ούτε από πλευράς ασφάλειας ούτε από τις ε, συνθήκες οδήγησης ε, με τη συμπερίληψη των αυτοαπασχολουμένων στο χρόνο εργασίας. Διότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο και υπέρ το δέον γραφειοκρατικό να ελέγχουμε και τον υπόλοιπο χρόνο πέραν του χρόνου οδήγησης για τους αυτοαποσχολούμενους οδηγούς. Υπάρχει και ένας μύθος που λέει ότι ο περιορισμός του χρόνου οδήγησης ε, είναι καλός ε, για την ασφάλεια, για την οδική ασφάλεια. Σαφώς δεν είναι κακός για την οδική ασφάλεια, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Τα βαρέα φορτηγά οχήματα πολλές φορές συμμετέχουν σε ατυχήματα σε ποσοστό 6% που σημαίνει ότι για όλα τα ατυχήματα που έχουμε το 6% περιλαμβάνουν και βαρέα φορτηγά οχήματα. Και το 16% είναι θανάσιμα ατυχήματα. Αλλά αυτό είναι συμμετοχή, δεν είναι ευθύνη του οδηγού το ποσοστό ευθύνη των οδηγών φορτηγών οχημάτων για τα ατυχήματα είναι κάτω του 6% για τα γενικά ατυχήματα, κάτω του 16% για τα θανατηφόρα ατυχήματα και νομίζω ότι με βάση τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε είναι καλά τα στοιχεία αυτά και δεν ισχύει να λέμε ότι μία σειρά από μελέτες επιβεβαίωσαν ένα τέτοιο θέμα. Δεν ισχύει να λέμε ότι οι οδηγοί φορτηγών οχημάτων αποτελούν δυσανάλογο αριθμό οδηγών για την οδική ασφάλεια είναι το ίδιο καλή ή κακή με οποιονδήποτε άλλο οδηγό. Μπορεί να είναι και καλύτερη γιατί έχουν πολύ καλύτερε επαγγελματικέ ε, δεξιότητες από άλλους οδηγούς. Κύριε Λίχτεμπέργκερ, ισχύει αυτό που σας λέω, βασίζεται σε ε, στατιστικά στοιχεία. Το θέμα όμως εδώ είναι να λέμε σαφώς ποιος καλύπτεται και ποιος δεν καλύπτεται από αυτή την οδηγία. Γι' αυτό ακριβώς και φροντίσαμε ιδιαίτερα το θέμα του καθορισμού των εργαζομένων αυτών όλων που βρίσκονται στο περιθώριο των ορισμών, στα όρια των ορισμών και ε, με πιο ελαστική ερμηνεία της οδηγίας μέχρι τούδε έχει αποκλειστεί από τον ορισμό, ενώ στην πράξη πρόκειται για υπαλλήλου, για απασχολούμενους εργαζομένους, γιατί ακόμα και αν δεν έχουν μια επίσημη σύμβαση εργασίας με έναν εργοδότη, στην πράξη συνεργάζονται με έναν μόνο αποστολέα, με, με μία μόνο μεταφορική εταιρεία και το αποκλειστικό, το σύνολο του εισοδήματός τους ε, εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τα όσα λαμβάνουν ως μισθό από αυτή την επιχείρηση. Και αυτοί οι οδηγοί φορτηγών οχημάτων είτε περιγράφονται ως ε, αυτοαπασχολούμενοι είτε ως υπάλληλοι βάσει της νομοθεσίες πρόκειται για υπαλλήλους, για απασχολούμενους ε, εργαζομένους, επομένως θα πρέπει να εμπίπτουν στο πλαίσιο της οδηγίας για να διασφαλίζονται τα εργασιακά τους δικαιώματα αλλά και η υγειοδική ασφάλεια. Αυτή είναι η πρόταση που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτή είναι και η αιτιολόγηση που δίνουμε. Θα ήθελα να προσθέσω ένα σημείο για την εκτερινή εργασία. Το υφιστάμενο κείμενο της οδηγίας όπως προέκυψε από τις δύσκολες διαπραγματεύσεις οι οποίες οδήγησαν τελικά στην υιοθέτησή του, καταλήγει να θεωρεί νακτερινή εργασία ακόμα και το παραμικρό λεπτό οδήγησης στις 4 ώρες, το διάστημα αυτών των 4 ωρών που τα κράτη-μέλη έχουν αποφασίσει ότι συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την εκτερινή εργασία. Αυτό δεν είναι λογικό, δεν είναι πρακτικό, δεν συνάδει με την κοινή λογική και δεν έχει να κάνει με την ειδική ασφάλεια. Θα πρέπει ε, να τακτοποιηθεί λίγο κάποιος αυτός ο κανόνας για να μπορεί να εφαρμοστεί. Γι' αυτό και ακριβώς προτείνουμε μία περίοδο δύο ωρών εντός αυτού του ορισμού της νύχτας που δίνεται από τα κράτη-μέλη να θεωρείται νεκτερινή εργασία και Έχω διαπιστώσει ότι υπάρχουν κάποιες τροπολογίες για να μειωθεί αυτό το χρονικό διάστημα. Είμαστε ανοιχτοί προ συζήτηση για το θέμα αυτό. Αυτό που έχει σημασία για μας είναι να έχουμε ένα λογικό ορισμό της νυχτερινής εργασίας που δεν μπορεί να θεωρεί το κάθε λεπτό οδήγηση ως νυχτερινή εργασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπλόκλαντ για να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σχετικά σύντομος, γιατί θα συμφωνήσω απόλυτα με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος όντως έδωσε κάποιες απαντήσεις τις οποίες θα ήθελα και εγώ να δώσω, πρώτου παρέχοντα το λόγο, να αναφέρω κάποια σημεία. Το πρόβλημα που ανέφερε ο κ. Γκρός για τα μεγάλα φορτηγά που ξεπερνούν τους 3,5 τόνους έναντι των μικρών φορτηγών κάτω από το όριο των 3,5 τόνων. Καταλαβαίνω το πρόβλημα, αλλά δεν βλέπω ότι μπορούμε να το λύσουμε στην παρούσα οδηγία. Με κάποιον άλλο τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Και νομίζω ότι έχουμε διάφορα να πούμε. Ωστόσο, κάθε όριο που θέτουμε είναι ένα, αν θέλετε, αυθαίρετο όριο για τον κύριο Κούστατσερ ανέφερε τα πολλαπλά ατυχήματα με τα φόρτιγα. Ναι, μα φυσικά κάθε ατύχημα είναι υπερβολικό. Είναι ένα ατύχημα το οποίο δεν θέλουμε να συμβεί και συμβαίνουν πολλά ατυχήματα με τα φόρτιγα. Δεν έχει αποδειχτεί όμως ότι αυτό απασχολούμενοι προκαλούν πιο πολλά ατυχήματα από τους μισθωτούς μιας εταιρείας και πολύ πιθανόν η εμπειρία των οδηγών να είναι τέτοια που όταν έχουν το δικό τους υλικό να συμπεριφέρονται καλύτερα και θα πρέπει φυσικά να έχουν και χρόνο για τα διοικητικά τους. Δεν βλέπω λοιπόν γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο συγκεκριμένο θέμα και επίσης γι' αυτό δημιουργήθηκε η οδηγία για την ανάπαυση. Εκεί θα λύσουμε τα προβλήματά μας. Δεν χρειάζεται εδώ στην οδηγία αυτή να το ρυθμίσουμε και σε δύο διαφορετικές οδηγίες να λύνουμε το ίδιο θέμα. Νομίζω ότι το πρόβλημα ε, επιλύεται σε ό,τι αφορά τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης και δεν χρειάζεται να εισαχθεί εδώ και πάλι το θέμα αυτό. Και φυσικά θα πρέπει στο επίκεντρο να είναι η οδική ασφάλεια, αλλά αυτό γίνεται ό,τι στην οδηγία για την ε, χρόνο χρονοδήγηση και ανάπαυσης. Για τον έλεγχο και την υποπτία τώρα, ναι, Όντως, οι αυτοπασχολούμενοι κάνουν τη δουλειά τους όσο θεωρούν ότι πρέπει να την κάνουν και αυτό δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Ο κύριος Βιασεμπόφσκι είπε ότι «Α, κι εγώ αυτοπασχολούμενος είμαι και δεν θέλω να έρθει κάποιος να με ελέγξει, να μου πει πόσο θα δουλέψω». Απόλυτα κατανοητό. Αυτό που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να το ελέγξουμε, να προσπαθήσουμε να το παρακολουθήσουμε, γιατί θα καταλήξουμε σε παταγώδη αποτυχία. Ποτέ δεν νομίζω ότι θα βρούμε νομοθεσία τέτοια και πού θα βρούμε τελικά κάποια νομοθεσία την οποία θα εφαρμόζουμε και θα παρακολουθούμε απόλυτα. Πρόεδρε, εδώ θα κλείσω και ελπίζω να ακολουθήσουν τον κατάλογο ψηφοφορία μου αύριο οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, πρωτού περάσω στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, θα ήθελα να σας επενθυμίσω ότι όλες οι εκθέσεις τις οποίες συζητούμε σήμερα θα ψηφιστούν αύριο. Ξεκινάει η ψηφοφορία στις 9 και 4. Εδώ στην αίθουσα αυτή αύριο το πρωί. Και να περάσω στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Στην πρόσβαση στην αγορά διεθνών οδικών... Συγγνώμη, πρόσβαση στην διεθνή αγορά μεταφορών με Πούλμα και λεωφορεία να δώσω το λόγο στον εισηγητή, στον κύριο Γκρός. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και ελεοφορία αλλά και των ε, εμπορευματικών μεταφορών νομίζω ότι μπορούμε να τα κοιτάξουμε μαζί αυτά τα θέματα. Να πω στους συναδέλφους ότι έχουν διοργανωθεί διάφορες συναντήσεις. Τρεις τεχνικές συναντήσεις διοργανώθηκαν τρεις ανεπίσημες ε, τριμερείς ε, συζητήσεις και με τους κοιόδης επίσης τρεις συναντήσεις και η κατάσταση είναι απλή αλλά όχι εύκολη. Να σας πω με απλά λόγια ότι όλη η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από δύο θέματα. Και ίσως το ένα να είναι αντίθετο με το άλλο σε ό,τι αφορά τα λεωφορεία, τη ρύθμιση των 12 ημερών και σε ό,τι αφορά τα εμπορεύματα, το καμποτάζ στα λεωφορεία. Να υπενθυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν την ψηφοφορία στην ε, Ολομέλεια εισήγε εκ νέου αυτή την ρύθμιση των 12 ημερών και ότι η κοινή θέση σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση των 12 ημερών δεν ελήφθη υπόψη. Αυτό σημαίνει επίσης αυτό σημαίνει επίσης ότι ζητήσαμε από το Ευρωπαϊκό ε, Συμβούλιο να μας πει αν ε, αποκλείονταν κάθε συζήτηση για το θέμα αυτό. Και το Συμβούλιο είπε ότι μια συμφωνία ITR που έχει ήδη υπογραφεί με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση της συζήτησης και ότι δεν ε, ήταν αποκλειστικά Δεν ήταν η βάση δηλαδή μόνο αυτή η ρύθμιση των 12 ημερών για το συμβιβασμό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πέραν τούτου, νομίζω ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά προβλήματα σε ό,τι αφορά τα λεωφορεία και τα πούλμαν. Θα ζητούσα απλά, αν ε, καταλήξουμε σε μια συμφωνία στα πλαίσια τριμερούς διαλόγου με το Συμβούλιο, η εφαρμογή για τις 12 ημέρες να μην γίνει τον ε, Απρίλιο του 2011 προκειμένου αυτό το απόσπασμα να εφαρμοστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί πρόκειται για μια κατάσταση η οποία θα πρέπει να διορθωθεί σε ό,τι αφορά τις εμπορευματικές μεταφορές για το καμποτάζ. Δεν είναι απλό το θέμα αυτό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πλειοψηφία τάχθηκε υπέρ του ανοίγματο του καμποτάζ αυτού κατά τα επόμενα τρία έτη, περιορισμό δηλαδή σε τρεις επιχειρήσεις καμποτάζ σε 7 ημέρες σε πρώτη φάση και μετά για ολοκληρωτικό άνοιγμα. Το Συμβούλιο δεν συμφωνεί πραγματικά. Το Συμβούλιο θέλει το καμποτάζ να περιορίζεται σε τρεις ε, ημέρες και θεωρεί ότι θα πρέπει να διεξάγει η μελέτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αναλύσει ενδεχομένως ε, αν είναι απαραίτητο να ανοιχτούν άλλο το θέμα του καμποτάζ. Τελεία και παύλα. Αυτό που κάπως με φοβίζει, για να το πω έτσι, είναι η κοινή θέση και η περίφημη λέξη προσωρινά είχαμε συμφωνήσει και αυτό αποτέλεσε βάση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι ακριβώς αυτό το προσωρινά είχε οδηγήσει ε, τα κράτη-μέλη στο να επινοήσουν διάφορες λύσεις γιατί κανείς τελικά δεν ήξερε τι επιτρεπόταν και τι όχι. Γι' αυτό εξακολουθώ να πιστεύω ότι αυτός ο όρος το προσωρινά, ανεξάρτητα με το τι θα γίνει με το καμποτάζ, θα πρέπει να οριστεί για να μην ε, αναζητούν και βρίσκουν προσωπικές λύσεις τα κράτη-μέλη για τις άλλες πτυχές τώρα. Δεν αναφέρονται άμεσα σε ό,τι αφορά την οδηγία και την απόσπαση για παράδειγμα. Άλλοι θεωρούν ότι είναι αυτονόητη η εφαρμογή της, άλλοι προτιμούν να μην τη συζητήσουν. Ε, δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι σωστό είναι να βρεθεί ένας συμβιβασμό χωρίς να αναφερθεί το θέμα αυτό για συνδυασμένες μεταφορές τώρα. Και αυτό αποτελεί πρόβλημα γιατί μια συγκεκριμένη οδηγία αποκλεί το καμποζάλα αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις ε, ορισμένα κράτη-μέλη γνωρίζουμε ότι αυτά που ρυθμίζονται δεν μπορούν να αλλάξουν σε άλλη οδηγία. Άρα αυτό θα συνεπάγεται προβλήματα. Γιατί πρόκειται και για τις χώρες αυτές οι οποίες πριν από κάποιους μήνες ήταν υπέρ της απελευθέρωσης των αγορών. Όντως, κάποιες χώρες επιδεικνύουν προστατευτισμικές τάσεις οι οποίες θεωρώ ότι είναι πολύ ανησυχητικές. Αν και πρόκειται για λεπτομέρεια, να σας πω ότι αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα ζητήσαμε μια συνοχή με, το, με την έκθεση της συναδέλφου Στικάου. Ελπίζω να πετύχουμε την χρονική αυτή συνοχή και να μην επισέλθουμε σε οι ημερομηνίε που ουσιαστικά, να σα θυμίσω και τι έγινε με την οδηγία για τα διπλώματα οδήγηση. κάποια προβλήματα λύθηκαν ουσιαστικά βιολογικά, όχι μέσω νομοθεσίας. Φυσικά θα πρέπει να επιληθούν τα προβλήματα εντό μια εύλογη προθεσμία ώστε να έχουν και χρόνο εφαρμογή στα κράτη-μέλη. Τώρα για το θέμα του καμποτάζ των ενδομεταφορών. Νομίζω ότι αυτό που προτείνει το Συμβούλιο για τρει ανταμεταφορές ε, το μήνα θα λυθούν τα θέματα, δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Θα πρέπει επίση να είμαστε, να έχουμε την εγγύηση, την εξασφάλιση ότι σε καμία περίπτωση δεν θα συμπεριληφθεί αυτός ο όρος ε, προσωρινά. Θα το δούμε αυτό από Μάρτιο-Απρίλιο, όταν θα ανοίξει η αγορά και κάποιες ε, μεταφορικές εταιρείες θα έρθουν προς τα εμάς από άλλες χώρες. Νομίζω ότι θα οργιάσουν οι φήμες σε κάποιες χώρες. Κάτι άλλο. Το θέμα είναι να, μεταφορ... να περιορίσουμε τις ανταμεταφορές γιατί φοβούμαστε ότι θα οδηγήσει σε ε, οικονομικό ή χρηματοπιστωτικό dumping. Από την άλλη πλευρά προβλέπουμε και μέτρα μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα καταπολεμήσουν αν θέλετε τις ε, εικονικές ε, τα μεταγκαταστάσεις και το ξέρω αυτό σε διαφορά και από τις εμπειρίες μου με το Βέλγιο. Οι εταιρείε αυτές που έχουν μόνο, αν θέλετε, μια εικονική έδρα, ένα γραμματοκιβώτιο σε μια χώρα. Αν όμως το Συμβούλιο αντιδρά με τόσο προστατευτικό τρόπο που θέλει να περιορίσει τόσο πολύ τις αλλά από την άλλη δεν ε, προβλέπει μέσα για την ε, καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, νομίζω ότι πρόκειται για μια σπάνια συνέπεια. Θα πρέπει λοιπόν να θέσουμε σωστά μηνύματα. Η αγορά θέλει να γνωρίζει τι θα αντιμετωπίσει στο μέλλον. Θα εξαρτάται από 27 διαφορετικές νομοθεσίες ή θα υπάρχει μια ενιαία νομοθεσία. Δεν τίθεται θέμα ασφάλειας. Μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να καταδείξει ευελιξία και στους δύο τομείς, αλλά νομίζω ότι περιμένει ένα σαφές μήνυμα από το Συμβούλιο, όχι να λέμε στο ένα ναι και στο άλλο όχι. Επειδή, για παράδειγμα, ε, η χύψη χώρα θεωρεί ότι ο τομέας των μεταφορών αποτελεί εθνικό τομέα. Αυτές θα ήταν οι παρατηρήσεις μου για τα θέματα αυτά. Νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε κοινή θέση. Ιδάλλως, ε, σε μια ευαίσθητη χρονική συγκυρία θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε ε, τις εκκλήσεις του τομέα. Θα μας φέρει και θα μας ρωτήσει ο κλάδος τι κάνατε για να επιλύσετε τα προβλήματα αυτά. Να πω επίσης ε, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα επαγγέλματα. Αυτό προβλέπεται για αύριο στην ημερήσια διάταξη, αλλά θεωρώ ότι σημαντικό θα ήταν να διευκρινίσουμε το θέμα των εικονικών αυτών ε, εδρών και κατά δεύτερον είναι σημαντικό να καταρτιστεί και ένα χρονοδιάγραμμα σε ό,τι αφορά την έκθεση Τικάου ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα που θα δώσει σωστό χρόνο και εύλογη προθεσμία τα κράτη-μέλη για να προετοιμαστούν, όχι όμως να δώσουμε παράταση 5-6 ετών χωρίς λόγο. Ιδάλλως θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και θα έρθει η χύψη χώρα και να μας πει «Α, κοιτάξτε, δεν, ε, είναι, δεν συμβαδίζει η βάση δεδομένων μας με τις άλλες βάσεις δεδομένων». Νομίζω ότι αυτό δεν θα ήταν ε, Σωστό. Και αυτό προβλέπετε για αύριο για την έκθεση ΤΙΚΑΟ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι διαδικαστικό. Είχα πει ότι θα γινόταν μια συζήτηση για τις α, α, διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές, ότι θα συζητούσαμε και τα δύο θέματα αυτά μαζί εμπορευματικές δηλαδή και μεταφορές με πούλμαν και λεωφορεία και θεωρώ ότι συμφωνείτε όλοι από όλες τις πολιτικές ομάδες. Λοιπόν, συζητάμε και τις δύο εκθέσεις μαζί, διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές και διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία. Ήθελα απλώ να το διευκρινίσω αυτό και εφόσον συμφωνείτε έτσι θα εργαστούμε. Τώρα, εκ μέρου των σαλιστών η κυρία Σαγιάλα Ινές παρακαλώ. Κυρία Γελασέντερ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Γκρός ε, για όλο το ενδιαφέρον και το γεγονός ότι είναι ανοιχτό στο διάλογο για αυτά τα δύο θέματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και όλο ένα αλλάζουν στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης. Ως προς το πρώτο θέμα των πούλμαν και των λοφορείων, νομίζω ότι στον άτυπο τίτλο την περασμένη εβδομάδα από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπήρχε περισσότερο ενδιαφέρον για να το λύσουμε από τις αμφιβολίες που εκφράστηκαν στο Συμβούλιο, δηλαδή τα όσα έχουν να κάνουν με την προηγούμενη συμφωνία. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε τα δύο θέματα και αυτό της κυρίας Τιτσάου ως ένα πακέτο, διότι εμείς φαίνεται να προχωράμε πολύ πιο γρήγορα. Φαίνεται ότι το Συμβούλιο διαπιστώνει ότι έχει κάποια προβλήματα και εμείς προχωρούμε με το χρονοδιάγραμμα και νομίζω ότι για το καμποτάζ, το οποίο εξακολουθεί να είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα του θέματος και θα είναι ένα στοιχείο του μέλλοντος, ε, δεν θα πρέπει να αποφασίσουμε τόσο γρήγορα. Το θέμα των 12 ημερών μου φαίνεται καλό. Ως παράδειγμα ε, για την ελαστικότητα υπάρχουν και κάποιες πτυχές οι οποίες θα πρέπει να λάβουν ε, με υπόψη και οι κοινωνικές πτυχές έχουν προκύψει στο Συμβούλιο. Εμείς ε, θα θέλαμε να προχωρήσουμε με βάση την πρόταση του εισηγητή. Η πρόταση αυτή, αν θέλετε, ήταν ε, η μία πάνω στην άλλη, ακόμα και στην τελευταία φάση της ε, διαπραγμάτευσης, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για την ελαστικότητα όλου του τομέα. Η πλευρά των εμπορευμάτων φαίνεται ότι ήταν πολύ πιο ευαίσθητη ε, από τον ε, τουρισμό στις Άλπεις και άλλα θέματα. Όσον αφορά τώρα στο καμποτάζ, δεδομένου ότι τα προβλήματα στο Συμβούλιο είναι πιο περίπλοκα και δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, Εμπιστεύομαι πάρα πολύ τον εισηγητή και ελπίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσει να προσπαθήσει να βρει την άγουσα μέσω της οποίας θα μπορέσει να πείσει το Συμβούλιο ότι θα πρέπει να υπάρχει νομική ασφάλεια και ότι αυτά ε, τα θέματα των προθεσμών θα πρέπει να είναι σαφή. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τις αποφάσεις. Ε, μπορούμε να παραπέμψουμε και πάλι στις ελληνικές καλένδες το θέμα, ε, διότι φαίνεται, όπως μας λέει ο κλάδος, ότι έχουμε περιπλέξει την όλη κατάσταση του καμποτάζ με όλους τους υπολογισμούς που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή και ε, δεν φαίνεται να τους δίνουμε ένα σαφές μέλλον ε, για τον καθορισμό ενός κοινού χώρου για την μεταφορά εμπορευμάτων. Η ομάδα μου συζητάει και το θέμα των εργαζομένων σε υπηρεσίες ε, και ε, τον κοινωνικό αλλά και φορολογικό αντίκτυπο και πιστεύω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Συμβούλιο θα πρέπει να μας διασφαλίσουν ότι τα θέματα που τους θέτουμε και το τελικό αποτέλεσμα θα λάβουν υπόψη τους αυτές τις πτυχές έτσι ώστε να έχουμε νομική ασφάλεια αλλά και κοινωνική ασφάλεια και φορολογικές διασφαλίσεις. Τώρα, ως προς τα χρονοδιαγράμματα, συμφωνώ ότι θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι θα πρέπει να έχουμε μία περίοδο ε, θα έχουμε μάλλον μια περίοδο ε, αδράνειας λόγω των ευρωεκλογών και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη με αυτό διότι το θέμα μπορεί να πρέπει να συνεχίσει και μετά από τις εκλογές. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ο κύριος Στέρξ ε, θέλει το λόγο από πλευρά των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα ασφαλώς να σας ευχαριστήσω για αυτά που είπατε και το έργο σας. Τρία σημεία νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Μιλήσατε για προστατευτισμό και εσείς ο ίδιος και ο προστατευτισμός δεν περιορίζεται. Νομίζω ότι η ενιαία αγορά έχει συμφέρον να περιορίσει όσο το δυνατόν γίνεται το καμποτάζ. Κατά δεύτερον, Νομίζω ότι υπάρχει και μια περιβαλλοντική πτυχή στο έργο μας, γιατί θα πρέπει να περιοριστεί το καμποτάζ για το περιβάλλον, σε ό,τι αφορά το περιβάλλον. Τρίτο θέμα. Ε, αυτά που θα υποβάλουμε ως πρόταση θα πρέπει να είναι εφαρμόσιμα, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση ο μεταφορέας τελικά δεν καταλαβαίνει τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να τιμωρηθεί και το καθεξής. Νομίζω ότι αυτό που πρότεινε το Συμβούλιο δεν κινείται προς τη δική μας κατεύθυνση. Εγώ ήθελα να πάμε πιο πέρα από αυτά που πρότεινε και το Κοινοβούλιο και νομίζω ότι στα τρία σημεία αυτά δεν υπάρχει αποτέλεσμα αποδεκτό για μας. Νομίζω ότι στις διαπραγματεύσεις μας λοιπόν θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση. Εγώ θεωρώ ότι δύσκολα θα καταφέρω να συμφωνήσω γιατί η υφιστάμενη ρύθμιση μάλλον καλύτερη και η σημερινή ασάφεια παρά να δημιουργήσουμε μια τέτοια σαφήνεια. Να δημιουργήσουμε τέτοιους κανόνες που δεν ε, λειτουργούν. Νομίζω ότι θα πρέπει να επανέλθουμε λοιπόν στην τροπολογία 18 και να μειώσουμε τις περιορισμούς όπως είπε και ο Ματίας με με μια πλήρως ανοιχτή αγορά το 2014. Νομίζω ότι τα κράτη-μέλη μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν βρει ένα σύστημα για την ε, καταπολέμηση των εικονικών εδρών των εταιριών. Νομίζω ότι μπορούν να συζητούν τα κράτη-μέλη μεταξύ τους και ότι θα είναι απλή η συνεργασία τους αν υπάρχει η ανάλογη βούληση. Δεν θα πρέπει να αποδεχτούμε σε καμία περίπτωση ένα φορτηγό να πρέπει να διάζει τελείως προτού μπορεί να προβεί σε καμποτάζ. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ επιζήμιο. Και νομίζω ότι η όλη ρύθμιση που προτείνει το Συμβούλιο για τη διαμετακόμιση και την επιστροφή είναι πάρα πολύ περίπλοκη και ούτε καν εφαρμόσιμη. Νομίζω λοιπόν ότι θα, πούμε, θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να πρέπει να ακολουθείται ο η πιο βραχία απόσταση, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να επιβάλλουμε τα τρία καμποτάζ. Δεν νομίζω ότι είναι καλή λύση αυτή. Και νομίζω ότι όπου είναι δυνατή η συζήτηση και η συμφωνία, η σύναψη συμφωνία μεταξύ δύο κρατών μελών θα πρέπει να επιτρέπεται αυτό, γιατί και στους σειροδρόμους έχουμε συμφωνήσει ζητήματα, αν θέλετε, βάσει της αμοιβαιότητας. Δηλαδή ότι ανοίγει μια χώρα την αγορά της για κάποια άλλη, αν υπάρχει και η αμοιβαία σχετική ρύθμιση. Και νομίζω ότι και εδώ θα πρέπει να είναι δυνατό αυτό. Τα σημαντικότερα λοιπόν θέματα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για το ανοίγμα της αγοράς. Και μπορούμε να βρούμε και μέτρα, γιατί δεν είμαι υπέρ του χρηματοπιστωτικού dumping καθόλου. Αλλά δεν λέω ότι το άνοιγμα της αγοράς αυτόματα συνεπάγεται κοινωνικό dumping. Κατά δεύτερον, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται το καμποτάς και θα πρέπει να υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών που επιθυμούν να προβούν σε διμερείς ε, συμφωνίες. Νομίζω ότι θα πρέπει να τηρήσει σκληρή στάση ο εισηγητής και να μην υποχωρήσει ένα του Συμβουλίου. Ε, ε, Ευχαριστούμε πολύ. Μισή προτασούλα. Μισή σε ό,τι αφορά τις 12 ημέρες ο εισηγητής. Πραγματικά συμφωνώ απόλυτα με τον εισηγητή και αυτόν τον υποστηρίξω απόλυτα. Η κυρία να ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω στο θέμα αυτό για αυτά που ανέφερε και ο συνάδελφο Στέρεξ, ότι συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Το ελπίζω, λέει ο κύριο Στέρεξ. Γιατί στην αγορά αυτή το θέμα είναι και μιλώ σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση του καμποτάζ. Πολύ απλά οι καταστάσεις και οι συνθήκες στην Ευρώπη δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμες. Πώς να το κάνουμε. Ο αρνητικός αντίκτυπος σε διάφορες χώρες είναι διαφορετικού επίπεδου. Και αυτό έχει να κάνει σε πολλές περιπτώσεις και με θέματα απόστασης. Κάτι που σπάνια λέω, πρέπει να πω ότι κατανοώ κατά κάποιο τρόπο κάποιες θέσεις του Συμβουλίου και το γεγονός ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Το καταλαβαίνω αυτό τώρα, να λάβω θέση για κάποια θέματα σε ό,τι αφορά τα άδεια φορτηγά, σε ό,τι αφορά το καμποτάζ. Φυσικά και αυτό σχετίζεται με μία από τις βασικές υποθέσεις που μας απασχόλησαν. Κάποια στοιχεία που περιγράφονται ως καμποτάζ αν κάποιος φόρτωνε να κασώνει ντομάτες, αυτό έδινε δικαιώματα για καποτάζ στο κράτος μέλος της έντρας ή όχι. Αυτό είναι ένα αντικείμενο το οποίο έχει τύχει πολλών ε, καταχρήσεων. Λέμε ότι θέλουμε να αποφύγουμε το κοινωνικό dumping, αλλά θα ήθελα να υποδείξω και να σας καλέσω τα κράτη-μέλη να λάβουν υπόψη τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί και θα δούνε ότι υπάρχει πραγματικά τεράστια ποικιλία σε ό,τι αφορά τις κατάχρηση των κοινωνικών συστημάτων στην Ευρώπη. Υπάρχουν κατασκευές, αν θέλετε, υποδομές, ε, συστήματα, τις οποίες κανείς άνθρωπος δεν θα μπορούσε να σκεφτεί. Συστήματα που έχουν δημιουργηθεί για να αποφευθούν κοινωνικές ρυθμίσεις. Και αυτό φυσικά θα πρέπει να υπάρχετε σε κάποιον έλεγχο, γιατί ο ανταγωνισμός λειτουργεί όταν υπάρχουν δικαιοί όροι. Όχι όμως όταν γίνεται συστηματική κατάχρηση των κοινωνικών αυτών όρων, χρειάζεται κάποια παρακολούθηση. Δεν μπορούμε να το γλιτώσουμε αυτό. τα κοινωνικά συστήματα τα οποία υφίστανται τεράστια πίεση σήμερα στην Ευρώπη, συνάδελφοι. Αν τα θέσουμε σε κίνδυνο τα κοινωνικά αυτά συστήματα λέγοντας ότι αυτό το κοινωνικό ντάμπινγκ α, ας επιτραπεί και μιλάμε για φόρους, εισφορές στα κοινωνικά συστήματα, ε, να μην μας κάνει εντύπωση αν προκύψουν συστηματικά προβλήματα και σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των συστημάτων αυτών. Δεν είμαστε εδώ συνδικάτο για τα φορτηγά. Είμαστε εδώ για να εξισορροπήσουμε τα διάφορα συμφέροντα, για να δημιουργήσουμε νομική ασφάλεια για τους μισθωτούς, για τους εργαζόμενους στον τομέα αυτό. Για να μπορέσουν να υπολογίζουν και να ξέρουν οι επιχειρήσεις τι τις περιμένει στο μέλλον. Όχι όμως να, για να έχουν πλέον εκτίματα και να συνεχίζουν να καταχράζονται κάποιες επιχειρήσεις στα συστήματα των εθνικών κρατών μελών. Αυτό είναι κάτι το οποίο πώς να το κάνουμε δεν με βρίσκει σύμφωνη και εδώ θα πρέπει να πετύχουμε συμφωνία, γιατί εδώ μιλάμε για την οδική ασφάλεια, τους δίκαιους όρους, τις μεταφορές και τις δίκαιους όρους για την εργατική σχέση. Κύριε Γιασεμπόφσκι, σας ε, προκαλώ βαρεμάρα ίσως, αλλά και οι μικρές επιχειρήσεις ε, που υφίστανται αν θέλετε τις συνέπειες από τις μεγάλες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις και από την στρέβλωση του ανταγωνισμού, αυτές οι επιχειρήσεις, κύριε Γιατζεμπόσκι, νοιάζονται. Μιλάμε για απίσχναση ρυθμίσεων, οι οποίες θα ήταν σημαντικές σε ό,τι αφορά την προστασία σε ορισμένους τομείς. Αυτό λοιπόν με απασχολεί πάρα πολύ. Έχουμε καταβάλει τεράστιους σκόπους για τις ρυθμίσεις αυτές. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να εφαρμόζονται και σωστά, να παρακολουθούνται σωστά, να υπάρχει σωστή εποπτεία για να πετύχουμε ακριβώς αυτό το οποίο είχαμε υπόψη μας όταν ξεκινήσαμε να εξετάζουμε το θέμα αυτό. Είτε μιλάμε για το καμποτάζ, είτε μιλάμε για τις 12 ημέρες, για τις 12 ημέρες για τη σχετική ρύθμιση. Ναι, ασκήσαμε πίεση προκειμένου να καταλήξουμε σε συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους. Αυτό δεν ήταν κακό, θεωρώ. Και ήταν καλή η συμφωνία η οποία αποτύπωσε διάφορα συμφέροντα διαφόρων μέρων. Αν δεν είχαμε επιμείνει εμείς, δεν θα είχε προκύψει τίποτα. Μην τα αγνοείτε λοιπόν όλα αυτά και τα θεωρείτε γελία. Μιλάμε για τους δίκαιους όρους στον ανταγωνισμό. Αυτό θα πρέπει να αποκαταστήσουμε εδώ στις δύο αυτές ρυθμίσεις. Να είναι ξεκάθαρο αυτό. Εγώ δεν αδιαφορώ για τις δύο ρυθμίσεις και γι' αυτό τις εξετάζω τόσο λεπτομερώς. Κύριε Γαζεμπόφσκ, παρακαλώ. Συνάδελφε, αυτά που είπατε ωραία και καλά είναι, αλλά τι έχουν να κάνουν με το προκειμένο θέμα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Γερμανία, τουλάχιστον να ρωτήσετε τον κύριο Κράμαρε, θα διαπιστώσω ότι είναι ομοσπονδιακό κράτος και μέρο τη ενιαίας αγορά, Ωστόσο, η μισθή στη Φραγκφούρτη για τους εργαζομένου είναι πολύ διαφορετική, γιατί είναι διαφορετικέ και οι συνθήκες διαβίωση σε σχέση Φραγκφούρτη, μεταξύ Φραγκφούρτης και Μονάχου και Ζάρλαντ, είναι διαφορετικά τα ενίκια, ε, άρα είναι διαφορετική και η μισθή. Σε μία αγορά είναι διαφορετική η μισθή. Αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε είναι να υπάρχουν τεράστιε ε, διαφορές, αλλά είναι παράλογο να φανταζόμαστε ότι θα, θα, θα υπάρχουν μισθοί σε ένα και μόνο επίπεδο. Στη Γερμανία ακούμε για παράδειγμα ότι θα πρέπει να είναι παντού ίδιες οι συνθήκες διαβίωσης. Ωστόσο, επειδή διαφέρουν τα ενίκια στο Ούσμου και από το Μόναχο, για παράδειγμα, ή από τη Φραγκφούρτη, και αυτό διαφέρουν και οι μισθοί. Και στην Πορτογαλία φαντάζομαι ότι υπάρχουν ε, διαφορές μεταξύ Λισαβόνας και Πόρτο. Δεν είμαι κατά να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε την κοινωνική κατάχρηση. Είμαι υπέρ, αλλά αυτά τα αποκύματα πια της φαντασίας με κουράζουν. Να λέτε ότι, θέλετε, αλλά εμένα με κουράζουν για το καμποτάζ το καποτάζ αναλογεί σε 4% του συνολικού όγκου των μεταφορών. 4%. Είτε έχουμε λοιπόν ενιαία αγορά είτε δεν έχουμε. Φυσικά υπήρχαν μεγάλες διαφορές και είχαμε το ίδιο πρόβλημα και στη Γερμανία με τους βούλγαρους οδηγούς. Αν όμως πάντα λέω ότι α, υπάρχουν διαφορές και προσέχω τις παραμικρές λεπτομέρειες, ε, Στρεβλώνω την αγορά και αυτό δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε την κατάσταση, Ποιε ήταν οι διαφορές ε, στο συνθήκε διαβίωση ε, και στους μυθού του δεκαετία του 80, του 90, το 95, το 2000, το 2009 διαπιστώνουμε ότι σημειώθηκε αλλαγή. η μισθοί πλησιάζουν τα ίδια επίπεδα. Αλλά τι να κάνουμε, ξέρουμε ότι κάθε χώρα έχει διαφορετικό κοινωνικό σύστημα. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι οι Δανείοι ε, χρηματοδοτούν το κοινωνικό του σύστημα μέσω του ΦΠΑ. Οι Γερμανοί το κάνουν διαφορετικά. Ας μην λοιπόν υπερβάλλουμε. Υπάρχουν διαφορές, θα πρέπει να διαπιστώσουμε, να προσέχουμε, να ελέγχουμε ότι δεν υπάρχουν εξωφρενικέ διαφορέ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσουμε την ρύθμιση του καμποτάζ. Αποφασίσαμε με συντριπτική πλειοψηφία το 2014, το 2014, ενέτη 2009, έτσι. Η ρύθμιση του καμποτάζ η οποία ως σκόπο έχει να προστατεύσει με προστατευτικά μέτρα τους οδηγούς των φορτηγών να πάψει. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει και το 2018. Λέει όμως το Συμβούλιο ότι δεν θέλουμε ενιαία αγορά. Θέλουμε να προστατεύσουμε τους εθνικούς οδηγούς μας. Έμα ε, αυτό δεν αποτελεί ευρωπαϊκή προσέγγιση. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ και το λέω αυτό προς τον εισηγητή θέλω να πω δύο στοιχεία καταρχάς. Θέλουμε να, να υπάρχει όντω μια συμφωνία μεταξύ των θεμάτων και των εκθέσεων Gross Όχι όμως με οποιοδήποτε αντίτιμο. Δεν μπορώ να πω στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι θα παραμείνουν ε, οι περιορισμοί ε, για το καμποτάζ και θα κάνετε πίσω σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις για τα πούλμαν. Μπορούμε να και είμαστε διτεθειμένοι να κάνουμε πολιτικούς συμβιβασμούς, αλλά δεν μπορούμε να αποδυναμώσουμε τη ρύθμιση των 12 ημερών, γιατί αυτό που αποφασίσαμε και συμφωνώ κύριε Λεχτεμπέργκερ, ήταν η τελευταία αυτή η συμφωνία αποτέλεσε απόρρια των συμφωνιών με τους κοινωνικούς εταίρους και βλέπω ότι υπάρχει και διάθεση βελτίωσης από το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά το ΚΑΜΠΟΤΑΣ. δεν ε, μιλώ για το 2014 εδώ μπορώ να επιδείξω ευελεξία αλλά τώρα το να καθιερωθεί αυτό το προστατευτικό μέτρο στην ενιαία αγορά νομίζω ότι αυτό δεν μας επιτρέπεται ματιό και σε εμπιστεύομαι με την βελγική δεξιότητα, γιατί οι Βέλγοι είναι πολύ επιδέξιοι, ιδάλλως δεν θα υπήρχε πλέον το Βέλγιο καν, ε, σε εμπιστεύομαι λοιπόν και θα πρέπει όμως να σε ενισχύσουμε. Να πούμε ότι ναι, εντάξει, συμφωνία, αλλά όχι με κάθε αντίτιμο. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα που μπορούμε να αποστείλουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε την πρώτη αυτή φάση της συζήτησης, θα ακούσουμε τον κύριο Σίμψον. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω προσωπώντας αστικά μόνο τον εαυτό μου για την ομάδα την εκπροσώπηση η κυρία Γιάλα Σέντερ. Καταλαβαίνω λοιπόν ποια είναι η θέση του Συμβουλίου και υπό ποιε συνθήκε έχει καταλήξει μια θέση στο Συμβούλιο. Πιστεύω ότι όντω θα πρέπει να μπούμε στι πραγματεύσεις και να δούμε τελικά ποιο, ποια θα είναι η απόρριτη των πραγματεύσεων αυτών, αλλά καταλαβαίνω ότι ο χρόνο είναι πολύ σημαντικό στην πολιτική και το να υποβάλουμε τώρα την πρόταση αυτή, το να συζητάμε την πρόταση αυτή Πρώτον, σε μια φάση οικονομικής ύφεσης που δεν έχουμε δει εδώ και πάρα πολύ καιρό και λίγο πριν μάλιστα τις ευρωπαϊκές εκλογές θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα ατυχές. Και αυτό φοβάμαι ότι προς τα έξω θα δοθεί εντύπωση μια αρνητική μάλλον εντύπωση, γιατί καταλαβαίνετε ότι στα πλαίσια μιας προεκλογικής εκστρατείας ενώπιση των εκλογών τον Ιούνιο, όταν μιλάτε στον Ευρωπαίο πολίτη, οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για το καποτάζ, δεν καταλαβαίνουν καν τι θα πει η λέξη αυτή. Αυτό που τους ενδιαφέρει όμως είναι για ποιο λόγο θα επιστρέψουμε σε ξένους οδηγούς να κάνουν τόσα πολλά ταξίδια στη δική μας τη χώρα, όταν έχουμε τους δικούς μας οδηγούς φορτηγών, οι οποίοι με δυσκολία τα βγάζουν πέρα, με δυσκολία καταφέρουν να κάνουν τη δουλειά τους. Έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το είδαμε αυτό πριν από δύο εβδομάδες στον Ηνωμένο Βασίλειο με τους εργαζόμενους που εργάζονται στα δηληστήρια και σας διαβεβαιώ ότι δεν θα είναι μόνο οι Βρετανοί οι οποίοι θα αντιδράσουν γιατί όλοι θα νιώσουν πολύ άσχημα, πολύ σύντομα την ύφεση αυτή. Δεν μπορώ εγώ να πάω στους ε, οδηγούς φορτηγών της δικής μου χώρας, της δικής μου Πορτογαλ... Ε, εκλογικής περιφέρειας και να τους πω μην ανησυχείτε, τη δουλειά σας θα την κάνουν πλέον Ρουμάνοι και Βουλγα αλλά όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς και στα πλαίσια της εφαρμογής του κανόνα για το καμποτάζ. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε με αυτόν τον τρόπο στους Ευρωπαίους πολίτες. Και καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα έχουμε κάποια σημαντικά ζητήματα τα οποία πρέπει να επιλύσουμε. Από ό,τι φαίνεται δημιουργούμε μία σημαία ευκαιρία, αν θέλετε, εδώ πέρα, όπου υπάρχουν οδηγοί οι οποίοι νιολογούν εντό εισαγωγικών το φορτηγό του σε μία χώρα, δραστηριοποιούνται όμω σε μία άλλη και τελικά κερδοφορούν χωρί να καταβάλουν πουθενά φόρου. Όντω μπορεί τα συστήματα ασφαλείας, τα συστήματα ασφαλείας μπορεί κοινωνική ασφάλεια στα κράτη-μέλη να συγκλίνουν, σε καμία περίπτωση όμω δεν έχουν συγκλίνει πλήρω. Οι τιμέ επίση δεν έχουν ενερμανωστεί Και καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα δίκαιο επίπεδο ανταγωνισμού για όλους. παρόλα αυτά όμως, μόλον ότι δεν, έχουν, ε, δεν υπάρχουν ακόμα οι κατάλληλες συνθήκες, θέλετε εσείς να δημιουργήσετε ένα κλίμα εναρμόνισης, θέλετε να δημιουργήσετε κοινούς κανόνες για τον καποτάζ, χωρίς όμως να συνειδητοποιείτε ότι θα έχετε πάρα πολύ αρνητικές επιπτώσεις σε όλα τα κράτη-μέλη μέσω των κανόνων αυτών και χωρίς τελικά να λαμβάνετε υπόψη σας την ίδια την αντίδραση και την ίδια τη γνώμη των ανθρώπων που μας ψηφίζουν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή τη γνώμη των Ευρωπαίων πολιτών. Και αυτό που έγινε πριν από μερικές εβδομάδες στο Μένο Βασίλειο, στους εργαζόμενους δηλαδή για τη δίληση του πετρελαίου ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και κάτι το οποίο στιγμάτισε ουσιαστικά αν θέλετε την επικαιρότητα και το πρόβλημα δεν ήταν ότι ξαφνικά οι Βρετανοί στρέφονται εναντίον των ξένων εργαζομένων. Το πραγματικό ζήτημα και το, το πραγματικό αίτημα θέλει των ανθρώπων αυτών ήταν ότι θέλανε να έχουν ίδιες συνθήκες και ίδιους κανόνες εργασίας με τους αλλοδαπούς εργαζόμενους στο Μένο Βασίλειο. Και φοβάμαι ότι τέτοια προβλήματα διακριτικής μεταχείρισης θα δημιουργηθούν και με την έκθεση αυτή. Θα δοθεί εντύπωση ότι αφήνουμε στου να εργαστούν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να επιτρέπουμε όμως την αντίστοιχη ελευθερία και στους ε, γηγενείς ε, εργαζόμενους, στους Ευρωπαίους δηλαδή πολίτες. Σαφώς θέλουμε τις ίδιες συνθήκες και τις ίδιες τις ευκαιρίες για όλους. Για να δημιουργηθούν όμως ίσες ευκαιρίες για όλους, θα πρέπει να υπάρχει και ένα ισότιμο πεδίο εργασίας. Το ισότιμο αυτό πεδίο εργασίας δεν υπάρχει ακόμα. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει και οι Γερμανοί και οι Αυστριακοί ε, ε, οδηγοί φορτηγών να μπορούν να ανταγωνιστούν και αυτοί επί ίσης βάσης με τους ε, οδηγούς από άλλες χώρες. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερος; Ναι, Αναφερθήκατε στις ε, διαφορές που υπάρχουν και στις ε, διαφορετικές πληρωμές που υπάρχουν στη Γερμανία και ανάμεσα στα διαφορετικά κρατήδια της Γερμανίας. Δεν γνωρίζω εγώ ποιες είναι οι διαφορές αυτές εφόσον υπάρχουν. Εγώ αυτό μπορώ να πω ότι στο Μένο Βασίλειο έχουμε συλλογικές συμβάσεις, εθνικές συλλογικές συμβάσεις, επομένως το δικό σας επιχείρημα δεν μπορεί να ισχύσει. Αυτό το οποίο πρέπει να πετύχουμε εδώ πέρα να, να δώσουμε το σωστό μήνυμα, να δώσουμε μια σωστή εντύπωση προς τα έξω. Και επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπα στην αρχή. Αν τα πάντα ήταν ιδανικά, αν αυτή τη στιγμή ζούσαμε μια περίοδο οικονομικής άνθησης, αν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση για οδηγού φορτηγών, τότε στην περίπτωση μόνο αυτή η έκθεση αυτή θα ήταν λογική. Αλλά δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Δεν ζούμε σε μια τέτοια περίοδο. Οι συνθήκε είναι τελώς διαφορετικέ. Σας καλώ λοιπόν, πάση θυσία, να είμαστε προσεκτικοί. Προσπαθούμε σε κάθε περίπτωση να απελευθερώσουμε, να απορριθμίσουμε την αγορά και κάθε φορά βέβαια καταλήγουμε σε μια πολύ μπερδεμένη κατάσταση και τα πράγματα οδηγούνται σε μια πλήρη αποτυχία. Το είδαμε αυτό και με τον τραπεζικό τομέα. Αυτό μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι ότι μπορώ να συμφωνήσω με τον Ματιού και ε, να δούμε τελικά πού θα καταλήξουν οι πραγματεύσει, αλλά μη θεωρείτε το Συμβούλιο είναι αφελές και ότι δεν γνωρίζει ε, τι λέει και ότι είναι εκτός ε, ή κατά της ε, εσωτερικής αγοράς, ενδεχομένως να είναι λίγο κατά της εσωτερικής αγοράς αυτή τη στιγμή και ενδεχομένως να έχουν και δίκιο. Ακριβώς επειδή έχουν συνειδητοποιήσει τα κράτη-μέλη ότι οι οδηγοί φορτηγών τους υποφέρουν πάρα πολύ. Και το τελευταίο το οποίο πρέπει να κάνουμε εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να επιδεινώσουμε την κατάσταση. Ε, Έχουμε λίγα λεπτά. Υπάρχουν δύο ακόμα άτομα που έχουν ζητήσει το λόγο. Κύριε Σίμψον, Μία ερώτηση στον εισηγητή. Μετά από τους υπόλοιπους δύο που έχουν ζητήσει το λόγο θα σας δώσω το λόγο. Δεν ξέρω αν θέλετε να μιλήσετε μετά από αυτούς ή τώρα. Okay. Καλά. Να θέσω την ερώτηση ή να μην τη θέσω. Πέστε την παρακαλώ. Η ερώτηση είναι για την τροπολογία 3. Έχετε Μία τροπολογία τρία για τα συνδυασμένα ταξίδια βάσει της οδηγίας του Συμβουλίου. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό το combined transport journeys, αυτά τα συνδυασμένα ταξίδια. Για παράδειγμα, ε, η διέλευση κάτω από τη μάχη και τα ferry boat θεωρούνται συνδυασμένες μεταφορές, τότε ε, αν όχι, τότε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο είναι εκτός. Ο κύριος Κράμερ, παρακαλώ. Κύριε Γιαζεμπόφσκι, είπατε για να δικαιολογήσετε τη θέση σας ότι χρειαζόμαστε νέα αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει να είναι οργανωμένη και δεν είναι οργανωμένη. Συμφωνώ και λέτε για ότι πρέπει να υπάρχει κοινή φορολογική βάση και κοινό πλαίσιο. Βλέπουμε ότι τα φορτηγά της Ισπανίας περνάνε από το Λουξεμβούργο, μετά πάνε από τη Γερμανία στην Πολωνία επειδή είναι πιο φθηνά τα πράγματα εκεί. Αυτό είναι τρελό. Και αυτό δεν αφήνεται μόνο στα φορολογικά συστήματα, αλλά αφορά και την εθνική πραγματικότητα. Μπορεί δεν θέλετε να τα αλλάξετε αυτά και το ίδιο ισχύει για τους μισθούς. Και δεν μιλάμε μόνο για τους μισθούς. Φυσικά υπάρχουν διαφορές και στο επίπεδο αυτό, αλλά υπάρχουν και αν θέλετε ε, εύρη διαφορών. Και αυτά πρέπει να Δεν θέλουμε να τα ρυθμίσουμε. Αυτές οι διαφορές που υπάρχουν στις τιμές, για παράδειγμα, των καυσίμων, όλα αυτά προέρχονται από τα κράτη-μέλη. Αν θέλετε λοιπόν τέτοια ενιαία διαμόρφωση, να δούμε τι έχετε να πείτε για το φορολογικό δίκαιο. Γιατί δεν είναι δίκαια τα πράγματα, έτσι όπως μας τα λέτε σήμερα. Ευχαριστώ και για να ολοκληρώσουμε ο κύριος Γερζεμπόφσκι για άλλη μια φορά. Κύριε Κράμερ, ακριβώς το ευαίσθητο σημείο θίξατε, γιατί αυτό ήθελα να πω στον κύριο Σίμψον. Μιλάει για ενιαίους όρους, αλλά η δική του κυβέρνηση είναι κατά κάθε φορολογική συναρμόνιση Και οι πιο υψηλές τιμές για τα σπρίτι είναι στην ε, Βρετανία. Εγώ πάντα ήμουν υπέρ της έννοιας φορολογικής εναρμόνισης, αλλά τα κράτη-μέλη έχουν συμφωνήσει ότι δεν επιθυμούν αυτό. Δεν υπάρχει λοιπόν οποιαδήποτε ελπίδα. Μπορεί λοιπόν τα εθνικά κράτη-μέλη να λένε ότι σε σημαντικά θέματα θα πρέπει να συμφωνήσουμε και μετά θα συμφωνήσουμε για τις διαφορές και μετά θα καταστρέψουμε την ενιαία αγορά. Με την επιχειρηματολογία αυτή θα ξεκινήσουμε να αλλάξουμε και τις αεροπορικές συνθήκες. Δηλαδή, στη Βρετανία θα επιτρέπονται μόνο οι αεροπορικές εταιρείες που είναι βρετανικές ή οι Γερμανοί θα λένε μόνο γερμανικά αεροπλάνα στους γερμανικούς αερολιμένες. Ή... Αυτά θα ισχύουν λοιπόν και σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών και θα κάνουμε βήματα προς τα πίσω σε ό,τι αφορά την ενιαία αγορά. Όχι λοιπόν. Αυτά είναι ιδίες. Αιδίες. Φυσικά η ενιαία χώρα έχει πάντα κάποια μειονεκτήματα. Ποτέ δεν υπάρχει απόλυτη ισότητα στη δική μου χώρα και ακόμα και ο κ. Κράμας θα το παραδεχτεί αυτό. Στη χώρα μας επιμένουμε οι εταίροι μας, τα συνδικάτα, να ορίζουν τους μισθούς. Οι μισθοί όμως δεν ορίζονται από κρατικό επίπεδο. Αν δεν ορίζονται όμως από κρατικό επίπεδο, δεν έχω δυνατότητα να πω ότι α, θα είναι ενιαίο το μισθολογικό επίπεδο. Αυτά είναι ιδίες. Φίλημα. Μπράιον Σίμψον, καταλαβαίνω ότι έχει και τον προεκλογικό σου αγώνα, αλλά το γεγονό, ότι καταργούμε, θέλεις να καταργήσει μάλλον τι αρχέ τη ενιαία αγορά να σου πω το εξή αν προχωρήσουμε με τις, ε, τα επιχειρήματα που προτάσεις, μπορούμε να ξεχάσουμε την εσωτερική, την ενιαία αγορά. Να ανοίξουμε τους σιδηροδρόμους, όχι. Οι το γαλλικό μεσοδομικό δίκτυο ανήκει μόνο στους Γάλλους. Να μην ε, έρθει κανένας Γερμανός, κανένας Ισπανός, όχι η Γαλλία για τους Γάλλους. Ε, δεν ξέρω δηλαδή τι έχει συμβεί. Νόμιζα ότι είχαμε προχωρήσει λίγο παραπέρα από το σημείο αυτό. Temos ainda mais eh, e Σας ευχαριστούμε πολύ, ο κύριος Κίρκοπ. Και ελπίζω ότι δεν θα μιλήσετε για πάρα πάρα πολύ ώρα, γιατί πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Πρέπει να το πληρώσουμε σύντομα. Θα είμαι πολύ σύντομος, κύριε Πρόεδρε. Έχασα, αν θέλετε, το πρώτο τμήμα της παρέμβασης του κύριου Σίμψον. Έχοντας ακούσει βέβαια το τέλος της ομιλίας του και τα όσα είπε στη συνέχεια ο Γκέορκ, θεωρώ ότι τα τρία τελευταία λεπτά τουλάχιστον δεν ήταν ε, πολύ κακά και δεν νομίζω ότι ο κύριο Σίμψον θα αποφεληθεί ιδιαίτερα τη συζήτηση αυτή στα πλαίσια τη προεκλογική εκστρατεία, γιατί νομίζω ότι στον Ηνωμένο Βασίλειο είναι λίγο παγιωμένε οι απόψει όσον αφορά τα όσα συζητάμε. Συμφωνώ με τον Γεώργος προ το ότι ε, υπάρχουν πάρα πολλοί υψηλοί φόρη στο Ηνωμένο Βασίλειο και δασμοί και αυτό είναι γελίο θα έλεγα. Θα έλεγα ότι ουσιαστικά αποδυναμώνουμε την ίδια την θέση μας, δυσκολεύουμε τα πράγματα για εμάς τους ίδιους. Εγώ κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να έχουμε ένα ε, πλήρω ισότιμο επίπεδο στην εσωτερική αγορά και πιστεύω ότι δεν το καταφέρουμε εξαιτία των δικών μα λαθών και εξαιτία πολλών προτάσεων που κάνουμε εμεί οι ίδιοι. Νομίζω ότι ο Μπράιαν θα πρέπει ίσω να επιστρέψει στη χώρα του και να ζητήσει, αν θέλει, από την ίδια την δικιά του κυβέρνηση, ήταν λίγο πιο ευγενική με τον κλάδο, με το βιομηχανικό κλάδο. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ όλους, λέει ο Πρόεδρος. Δίνω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Πασκουαρέλη. Euh, euh, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω επικοδομητικά και αισιόδοξα, λέγοντας ότι ε, πέρα από τις ε, συζητήσεις αυτές για το καμποτάζι, για άλλα ευαίσθητα θέματα των δύο αυτών προτάσεων, έχει ήδη γίνει μια πολύ σημαντική εργασία και έχει ολοκληρωθεί πολύ σημαντική εργασία επιτυχώς προκειμένου να καταφέρουμε να συγκλίνουμε περισσότερο τις θέσεις του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο προκειμένου να καταλήξουμε συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση σε ένα κείμενο το οποίο δεν θα αναφέρεται μόνο στο καμποτάζ ή μόνο στον κανόνα των 12 ημερών ή μόνο στο ζήτημα της εικονικής έδρας αλλά που θα έχει να κάνει με το σύνολο των κανόνων αυτών που ζητάνε τα κράτη-μέλη προκειμένου να έχουν μια πιο εναρμονισμένη βάση παντού στην Ευρώπη προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες ανταγωνισμού στην Ευρώπη και προκειμένου να επικαιροποιηθεί και να εξυγχρονιστεί τελικά ένα πλαίσιο το οποίο είναι πλέον πεπαλαιωμένο, ένα πλαίσιο εργασίας. Ήδη πρόταση έχει υποβληθεί εδώ και αρκετό καιρό, πρέπει λοιπόν σύντομα να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και καταλαβαίνετε ότι το χρονοδιάγραμμα του Κοινοβουλίου, οι εκλογές αλλά και το χρονοδιάγραμμα άλλων θεσμικών οργάνων καλούν για μια ταχεία εργασία αυτή τη στιγμή, πρέπει να ολοκληρώσουμε γρήγορα. Επίσης όλη η συζήτηση που έχει γίνει για την έκθεση της κυρίας Τικάου είναι μια συζήτηση αρκετά θεωρητική αυτή τη στιγμή, βάσει των πρακτικών, σε σχέση με τα πρακτικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε τώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της προκειμένου να καταφέρουμε να συμφωνήσουμε γρήγορα, ενδεχομένως τον Απρίλιο, βάσει του κειμένου που θα εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε επίπεδο Συμβουλίου πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε τον Ιούνιο. και πέρα από το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να δούμε τα ουσιαστικά ζητήματα που βέβαια είναι το καποτάζ και ο κανόνας των 12 ημερών όσον αφορά το πρώτο, το καποτάζ. Νομίζω ότι το εφιστάμενο κείμενο της κοινή θέσης αποτελεί μια σημαντική πρόοδο σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Το καποτάζ ως παροχή υπηρεσίας πέρα από τη χώρα εγκατάστασης είναι μια διαδικασία, είναι μια πράξη προσωρινή. Πρόκειται για έναν κανόνα της συνθήκης που ισχύει για όλες τις υπηρεσίες και για τις υπηρεσίες μεταφορών. Πρόκειται για μια προσωρινή υπηρεσία, είτε αυτό καταγράφεται ρητός ή όχι στο κείμενο. Και νομίζω ότι όλοι συντοποιούμε τι εννοούμε με τον όρο temporary, προσωρινό και πολλές φορές και αποφάσεις του ΔΕΚ δεν μας επέτρεψαν να προχωρήσουμε γρήγορα. Γι' αυτό το λόγο το Συμβούλιο κατέληξε σε μια ρεαλιστική πραγματιστική θέση, ενδεχομένως να υπάρχουν και καλύτερες λύσεις. Αποφάσισε πάντως ότι ε, η πλήρης απελευθέρωση του καμποτάζ δεν ανταποκρινόταν στα προβλήματα που ε, είχαν εντοπιστεί. Πέρα από άλλα προβλήματα που ενδεχομένω να είχαμε εντοπίσει, όπως για παράδειγμα η φορολογική νομοθεσία κτλ. Ποια είναι τώρα η άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ζήτημα αυτό. Πιστεύουμε ότι θα ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο και το λέω πραγματικά πολύ ειλικρινά, θα ήταν πολύ επικίνδυνο να ανοίξουμε πάλι το κοντέ τη Πανδώρας όσον αφορά την κοινή θέση. Ωστόσο κύριε Γερζεμπόφσκι, καταλαβαίνω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνειδητοποιεί ότι δεν πρόκειται για μια οριστική λύση και ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να βρούμε μια λύση και ότι θα πρέπει μέσα στο κείμενο και πέρα από την έκθεση ή την κοινή θέση που θα έχουμε για το 2013 θα πρέπει στο κείμενο να υπάρχει μια πιο ένα πιο δυνατό κίνητρο προκειμένου να καταλήξουμε σε μια γενικότερη εναρμόνιση των υπηρεσιών αυτών έτσι ώστε κάποια στιγμή να καταφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια ολοκληρωμένη πρόταση. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες που εξέφρασαν ο κύριος Σίμψον και άλλοι, ιδίως ε, την περίοδο αυτή, την περίοδο της ε, οικονομικής χρηματοπιστωτικής κρίσης που διανύουμε. Αλλά θα μπορούσε να εξηγήσει ο κύριος Σίμψον στους εκλογείς του ότι το καμποτάζ είναι ένα equal playing field για όλους. Γιατί όπως οι οδηγοί φορτηγών από τα άλλα κράτη-μέλη μπορούν να πάνε στο Ηνωμένο Βασίλειο για παροχή υπηρεσιών καμποτάζ, κατά τον ίδιο τρόπο και οι Βρετανοί οδηγοί φορτηγών βάσει των ίδιων ακριβώς κανόνων μπορούν να μεταβούν σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Υπηρετική Ευρώπη για παράδειγμα, για να παρέχουν υπηρεσίες καμποτάζ. Να πω επίσης ότι πρέπει να διευθετήσουμε και το ζήτημα των συνδυασμένων μεταφορών. Ουσιαστικά όμως πρόκειται για ένα εικονικό πρόβλημα. Δεν αποτελεί πρόβλημα το ζήτημα των συνδυασμένων μεταφορών. Το καμποτάζ είναι μία εθνική υπηρεσία, θέλετε. Δηλαδή ξεκινάει σε ένα άλλο κράτος μέλος που δεν είναι το κράτος μέλος ε, προέλευσης, ενώ οι συνδυασμένες μεταφορές από τη φύση τους είναι διεθνείς μεταφορές. Επομένως δεν υπάρχει λόγος να γίνεται σύγχυση ανάμεσα στις συνδυασμένες μεταφορές και τον καμποτάζ. Και αν με επιτρέπει ο κύριος Γκρός να απαντήσω στην ερώτηση που έθεσε ο κύριος Σίμψον, θα έλεγα ότι ε, η μεταφορά των φορτηγών στη μάχη είτε γίνεται μέσω του τούνελ, είτε γίνεται με ferry boat, δεν έχει να κάνει, δεν υπάγεται καθόλου στον ορισμό των συνδυασμένων μεταφορών. Και να αναφερθώ επίσης και στον κανόνα των 12 ημερών. Ο κανόνας αυτός βέβαια έχει να κάνει με τη μεταφορά, έχει να κάνει με τη μεταφορά επιβατών με πούλμαν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να υποστηρίξει την τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το κείμενο αυτό αποτελεί αποτέλεσμα συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προβλέπεται επίσης στα πλαίσια της συμφωνίας ΕΤΕΡ, την οποία θα καταφέρουμε να παρουσιάσουμε σύντομα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε λοιπόν πλέον στα χέρια μας ένα ρυθμιστικό κείμενο το οποίο συνάδει πλέον με την τροπολογία του κύριου Κρός την οποία μπορεί να υποστηρίξει βέβαια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι ε, κατά αυτόν τον τρόπο ε, διασκεδάζονται και ανησυχίες πολλών κρατών μελών που είχαν ε, θέσει ζήτημα διακινδύνευσης οδικής ασφάλειας μέσω του κανόνα των 12 ημερών. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι δεν θα έχουμε τον κανόνα των 12 ημερών που είχαμε σε παλαιότερους κανονισμούς πριν από το 2006. Έχουμε έναν νέο κανόνα πλέον των 12 ημερών, πολύ πιο συγκεκριμένο που λαμβάνει σαφώς υπόψη του το ζήτημα της οδικής ασφάλειας. Καταλαβαίνετε ότι μέσω του νέου κανόνα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών σε συνεχή βάση χωρίς να προβλέπεται χρόνος ανάπαυσης. Ευχαριστώ και για να τελειώσουμε τη συζήτηση ο λόγος στον εισηγητή. Ευχαριστώ πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Δεν θα ήθελα να ξαναξεκινήσουμε την όλη συζήτηση για την ενιαία αγορά. Νομίζω ότι και ο Μπράιν και ο Γκέορκ έκαναν ε, ό,τι μπορούσαν και έδωσαν τις καλύτερες συμβουλές για το θέμα αυτό. Η προσωπική μου ε, προσωπική άποψη θα παρέμενε στο θέμα της ερώτησης αν περιοριστούν οι δραστηριότητε σε, μια χώρα, αν αυτό κατά ανάγκη σημαίνει ότι ε, χρονικά στο μέλλον θα προκύψει πιο έντονη εναρμόνιση. Αυτό που έχω διαπιστώσει εγώ και νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν τις απόψεις μου Αυτό που διαπίστωσα λοιπόν εγώ είναι το εξής. Όπου τουλάχιστον σε διεθνές επίπεδο υπάρχει εντατική συνεργασία, η εναρμόνιση ερχόταν πιο γρήγορα από ότι σε αντίθετη περίπτωση. Και αυτό μπορεί να αποδειχτεί σε ό,τι αφορά την φορολογική πολιτική. Δυστυχώς το γεγονός ότι ένας ε, μισθωτός ε, βρίσκεται τακτικά σε κάποια άλλη χώρα δεν επηρεάζει την φορολογική πολιτική. Αν σε κάποιο χώρα στάθμευσης ε, συναντηθούν κάποιοι οδηγοί και συγκρίνουν τους μισθούς τους, αυτό γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Δεν ξέρω όμως ε, αν έχει σκοπό η εναρμόνιση αυτή. Αυτή λοιπόν η παρατήρησή μου να εξετάσουμε το θέμα αυτό εξ αρχής. Γι' αυτό που είπε ο Μπράιαν, δεν είναι ατυχής η χρονική συγκυρία και το χρονοδιάγραμμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το χρονοδιάγραμμα και ευτυχώς ε, εγκαίρος, ε, μάλλον όρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Ορών προσωρινά ιδάλως. Το 2009 θα είχαμε χώρες οι οποίες θα σκούσαν μέτρα καμποτάς και θα αντιμετώπιζαν διαφορετικές νομικές ρυθμίσεις σε κάθε χώρα. Είναι σημαντικό να το επεξεργαστούμε αυτό και δυστυχώς η Γαλλική Προεδρία δεν έδωσε προτεραιότητα στο θέμα αυτό. Ιδάλλως θα το είχαμε ολοκληρώσει το φθινόπωρο του 2008. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις προτάσεις, σου, για τις προτάσεις του. Και φυσικά με τις τροπολογίες μου ήθελα να υποδείξω κάποιες κατευθύνσεις και όπου δεν υπάρχει συμβαστική πρόταση θα ήθελα να επανέλθουμε ε, στην αρχική στάση του Κοινοβουλίου. Χαίρομαι που οι συνάδελφοι μου δώσαν κάποιο περιθώριο ελιγμού. Ξέρω ότι δεν είναι πρώτο θέμα και θα περιοριστούν, θεωρώ, οι συζητήσει στα δύο αυτά βασικά θέματα. Για τις λεπτομέρειες έχει συζητηθεί ήδη πάρα πολύ και θα ρυθμιστούν και από μόνες τους αν ρυθμιστούν τα δύο βασικά θέματα σε ό,τι αφορά το τρανζικ, καμποτάζ, τις ε, διμερείς, πολυμερείς συμφωνίες κτλ. Νομίζω ότι αν έχουν ρυθμιστεί τα δύο βασικά θέματα, να τα ξανακοιτάξουμε και αυτά. Θεωρώ ότι θα πρέπει τη ρύθμιση των 12 ημερών να τη διατηρήσουμε με ισόρροπη μορφή. Το καμποτάζ θα πρέπει να είναι σαφές και να μην εμείνουμε στον όρο προσωρινά. Αυτό δεν θα έχει αποτέλεσμα, θα βλάψει και τις χώρες και τις επιχειρήσεις και το Συμβούλιο θα πρέπει να μας δώσει ένα μήνυμα αναφορικά με την ενιαία αγορά και την ερμηνεία που της δίνουμε τα τελευταία 10 χρόνια και θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτό, αυτή η ενιαία αγορά θα πρέπει να ε, αφήνει περιθώρια και για κάποιες διαφορές οι οποίες σταδιακά θα επιληθούν. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, η συζήτηση ήταν μακροσκελέστατη. Νομίζω ότι πλέον διαθέτουμε μια κοινή βάση και στοιχεία πάνω στα οποία μπορούμε να στηρίξουμε τις θέσεις μας και να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συνένεση. Αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι οι προθεσμίες. Προθεσμία έχουμε 25 ε, Φεβρουαρίου 12 το μεσημέρι για κατάθεση τροπολογιών, ψηφοφορία στην Επιτροπή 31 Μαρτίου και στην Ολομέλεια του Απριλίου θα συζητηθώ το θέμα. Με αυτό νομίζω έχουμε ολοκληρώσει με την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης και τώρα έχουμε συνεδρίαση των συντονιστών. 5-10 λεπτάκια για να φύγουν όσοι δεν ε, έχουν ε, δουλειά και ευχαριστώ και τους ερμηνείς.